είπε η κυρία Άουκεν. Θέματα της κυρίας για τα οποία εν μέρει απήντησε ο Ισπανός κύριος. Έχουμε την καταγγελία που τόσε ήρθε σε σχέση με την παραβίαση του δικαιώματος της όπω όπως λένε οι αναφέροντες, το Κοινοβούλιο τα έχει συζητήσει αυτά στην Ολομέλεια. Οπότε το κοινοβούλιο βλέπετε ότι είναι κοινοβούλιο, ασχολείται πολιτικά, δεν ασχολείται σαν να είναι δικαστήριο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θα ήθελαν ίσως οι πολίτες αλλά και οι βουλευτές. Θα πρέπει να ασκήσουμε την πολιτική μας επιρροή με τέτοιο τρόπο που να επηρεάσουμε εθνικές, πολιτικές, τέλος πάντων τοπικές αρχές στα κράτη-μέλη και έτσι τελικά ίσως να επιτευχθεί η απόνομη δικαιοσύνη ει όφελο του αναφέροντο. Έτσι το βλέπουμε και γι' αυτό λοιπόν και μας λένε και τα δικά του, ε, όσοι έχουν να οι καλεσμένοι μας από αυτή τη θέσεως. ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο αυτής αμέσω στους προσκεκριμένους μας το και να έχουμε μετά το χρόνο τόσο ώστε να μπορούμε να κάνουμε εδώ απαντήσεις. Σαμπίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κατηγορία θεμελιωδών δικαιωμάτων α, παραπών θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ίσως είναι περίεργη αυτή η διατύπωση, αλλά να σας την εξηγήσω. Με βάση συνθήκη της Λισαβόνας έχουν, έχει ενσωματώσει η συνθήκη το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στις συνθήκες, αλλά δεν έχει δημιουργήσει ένα δικαίωμα δράση, ούτω ώστε να εφαρμοστεί ο, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό διαφέρει από αυτό που συνέβη με την αρχή της επικουρικότητας, όπου το δικαίωμα δράσης έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την αρχή αυτή. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, δυνατότητα καταγγελίας λόγω παραβίασης αυτού του θεμελιώδους δικαιωμάτου διοκαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου. Υπάρχει το δικαστήριο, το γενικό δικαστήριο και το δικαστήριο ε, δημόσιας διοίκησης. Οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται από τις συνθήκες και το καταστατικό του δικαστηρίου και για να ασχοληθούμε με, μια καταγγελία που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρχει υπόθεση μέσα στην ομολογία του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι σημαντικές υποθέσεις είναι αιτήματα για προδικαστικές αποφάσεις, όπου τα εθνικά δικαστήρια μπορεί να υποβάλουν ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ερμηνεία του, ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και για την ισχύ των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαδικασία προδικαστικών αποφάσεων είναι μια έκφραση αυτής της επικάλυψης που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, τη διασταύρωση ή της σχέσης μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως τα εγγυάται ο χάρτης που είναι δεσμευτικά για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και για τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο. Στην περίπτωση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη-μέλη φυσικά υπάρχουν και ένδικα ε, μέσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων αλλά για να γνωρίζουμε πώς θα ερμηνεύσουμε το χάρτη σε αυτές τις περιπτώσεις τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να αποτανθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για έκδοση προδικαστικών αποφάσεων. Μία άλλη σημαντική πτυχή των, ε, της δικαιοδοσίας των ε, ευρωπαϊκών ε, δικαστηρίων είναι η άμεση δράση από πολίτες εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όπως ξέρετε, αυτό το, το άμεσο δικαίωμα δράσης των πολιτών εναντίον πράξεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι αρκετά περιορισμένο. Γιατί το ενωσιακό δίκαιο στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά τους πολίτες μόνο μέσω των κατεφαρμογή του από τις εθνικές αρχές και όχι από τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρχει μια περίπτωση που φύγει ε, θεμελιώδη δικαιώματα, κάθε ένα από τα τρία δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, εξετάσει αν ισχύει ο χάρτης και αν ναι, να ερμηνεύσει και θα εφαρμόσει τις διατάξεις του χάρτη. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά σε περίπτωση α, καταγγελιών που δεν είναι αμυγός ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη ε, δράση για ακύρωση μια απόφαση ή ενό κανονισμού που υιοθέτησαν τα θεσμικά όργανα. Ε, υπάρχει μια έκκληση γιατί υπάρχει καταγγελία λόγω παραβίασης της συνθήκης κατά την εφαρμογή. Κατά την καταγγελία αυτή εξετάζουμε αν υπάρχει α, συνάφεια με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως είπε σήμερα το πρωί ο κύριο Νέμιτς, τα δικαστήρια έχουν συγκεκριμένο τρόπο να αντιμετωπίζουν αυτέ τι υποθέσει. Οι δράση μπορούν να πάρουν είναι συγκεκριμένοι. Υιοθετούν αποφάσεις ή εντολές. Και οι αποφάσεις που παίρνουν έχουν ε, επιπτώσεις. Μπορούν να ακυρώσουν πράξεις ή δράσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων οι αποφάσεις και εντολές αυτές ε, είναι εφαρμοστές, η ερμηνεία που δίδουν διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δεσμευτικές για τα εθνικά δικαστήρια που παρέπεμψαν ε, την υπόθεση και που έκαναν, υπέβαλαν το αίτημα. Η αρχή της ε, Αρμοδιότητα της δικαιοδοσιακή, όπως ανέφερε ο καθηγητής Ζακέ σήμερα το πρωί, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη η δικαιοδοσία και να μην υπάρχει ε, δυνατότητα να αποφασίσεις αν είναι δική σου υπόθεση ή όχι. Εάν υπάρχει μια υπόθεση λοιπόν και υπάρχει δικαιοδοσία, αν ισχύει ο χάρτη, τότε το δικαστήριο θα εξετάσει και θα εφαρμόσει το χάρτη αν υπάρχει μια υπόθεση χωρίς όμως δικαιοδοσία, τότε το δικαστήριο θα πάρει μια απόφαση και θα την ε, αιτιολογήσει. Αυτό έγινε σε διάφορες εντολές που εκδόθηκαν πρόσφατα για υποθέσεις που παραπέμφθηκαν τα εθνικά δικαστήρια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπό τη διαδικασία των προδικαστικών αποφάσεων, όπου τα εθνικά δικαστήρια ζήτησαν μία ερμηνεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κάποιων διατάξεων του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σε περιπτώσεις που εξέφευγαν του σκοπού εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Μην ξεχνάτε τι είπε σήμερα το πρωί ο καθηγητής της ΖΑΟΥ για την ανάγκη του καθηγητή Τεζάουρο να είμαστε εντός του πεδίου εφαρμογή του χάρτη, ο οποίος συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής του νοσιακού δικαίου. Αν εκφεύγουμε από το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύσει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα εξηγήσει το δικαστήριο γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί με μια υπόθεση και θα πει γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί ή θα πει ότι απαντώ στην ερώτηση που του τέθηκε, ε, σε περίπτωση όμως που έχει δικαιοδοσία, όπως είπα προηγουμένως. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί η αποστολή του είναι να αποφασίζει για υποθέσεις και όχι να δίνει νομικές συμβουλές. Επομένως, οι αποφάσεις των τριών δικαστηρίων δεν έχουν καμία ένδειξη, κανένα στοιχείο της παιδαγωγικού χαρακτήρα για εναλλακτικά ένδικα μέσα. Πέρα από τις υποθέσεις λοιπόν, τα τρία δικαστήρια φυσικά λαμβάνουν και πολυάριθμες επιστολές και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τους πολίτες που φύγουν θέματα πολύ διαφορετικά και επικοιλόμορφα μεταξύ τους και ορισμένα από αυτά αφορούν και θεμελιώδη δικαιώματα. Συνήθως αυτές οι επιστολές θα λάβουν μια απάντηση. Που είναι όμως τυποποιημένη απάντηση, που εξηγεί ποια είναι η δικαιοδοσία του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Και θα εξηγήσει γιατί το δικαστήριο δεν μπορεί να ασχοληθεί με τέτοιου είδους προβλήματα. Όταν είναι πολύ προφανής η υπόθεση, μπορεί να υπάρξει μια ένδειξη για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν παραπέμπουμε συστηματικά στους αρμόδιους φορείς. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Οπότε τώρα να δώσουμε το λόγο στον Βίκτορ, στο που εργάζεται στο Δικαστήριο των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ στην αρχιτεκτονική τη Ευρώπη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι το νομοθετικό σώμα με τη μεγαλύτερη ε, δικαιοδοσία και γιατί καλύπτει 27 κράτη-μέλη, γεωγραφικά δηλαδή, και σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή των διατάξεων που εφαρμόζει, τι διατάξει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή. Και σε αντίθεση με το χάρτη σημειώνουμε ότι η εφαρμογή της σύμβασης δεν περιορίζεται στον επιχειρησιακό, αν θέλετε, τομέα συγκεκριμένου δικαιικού συστήματος. Κάποια παραδείγματα, ας πούμε, που υπάρχουν στο έγγραφο μαζί με την έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή του χάρτη αναφέρεται ότι υποθέσεις σχετικά με μυστική παρακολούθηση ποινικές, στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών ή εθνικοποιημένης ε, ιδιοκτησίας δεν καλύπτονται. Αυτά όμως επηρεάζουν περιπτώσεις όπου που καλύπτονται από τη σύμβαση. Και το δικαστήριο έχει ε, εκδώσει σημαντικές αποφάσεις. Παράλληλα όμως η δικαιοδοσία του δικαστηρίου περιορίζεται από πολλές απόψεις, δεν καλύπτει κάποιες κατηγορίες όπως πολιτιστικά δικαιώματα καλύπτει μόνο πράξεις που αποδίδονται στις δημόσιες και κρατικές αρχές, όχι σε ιδιώτες. Και δεν επεκτείνεται για να καλύψει διακρατικά υπερεθνικά όργανα, ούτε επεκτείνεται πέρα από τα ενωσιακά ε, στα όργανα αφού προς το παρόν δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση η Ένωση. Σύντομα τώρα θα σας δώσω μια ιδέα για τους τομείς όπου και η σύμβαση και ο χάρτης μπορεί να ισχύουν και τους άλλους τομείς διαμορφώνεται η εξή εικόνα. Όταν υπάρχει θέμα θεμελιώδους δικαιώματος στην Ευρώπη, αν θέσουμε το ερώτημα με ποιο είναι ο αρμόδιος δικαστής, εκεί μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ τριών περιπτώσεων. Υπάρχει μια περίπτωση όπου δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο, και το ενωσιακό και σε αυτή την περίπτωση η εθνικοί φορείς και τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια. Αν καλύπτεται το θέμα από τις διατάξεις σύμβασης, μετά την εξάντληση των εθνικών ενδίκων μέσων μπορεί το πρόσωπο να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Και τέλος, περιπτώσει όπου εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Μπορεί δηλαδή τα ενωσιακά όργανα και φορείς να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το, Ευρωπα... το ε, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκείνο το δικαστήριο θα είναι αρμόδιο, εφαρμόζοντας πάνω απ' όλα το χάρτη, να κρίνει το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο δε χάρτης πρέπει να ερμηνευθεί και στο φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και της νομολογίας για του δικαστηρίου. Εδώ σταματάει η απαρίθμηση. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι μπορεί να ξεπεραστεί η συνθήκη αυτή και μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να ε, παρεμβαίνει και το δικαστήριο του Στρασβούργου. Σε άλλη περίπτωση όπου εφαρμόζεται το δίκαιο και όπου τα εθνικά δικαστήρια λειτουργούν, τότε η διαδικασία στη συνέχεια που θα δοθεί είναι σε τοπικό επίπεδο να εξεταστεί η διαφορά, να εξεταστούν και τα θέματα ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων και μετά τα δικαστήρια, αν εφαρμόζεται ο ενωσιακό δίκαιο, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα δικαστήρια και το χάρτη και τη σύμβαση. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ή μάλλον η δυνατότητα να υπάρχει ε, προδικαστική απόφαση όπου το δικαστήριο θα ερμηνεύσει το ενωσιακό δίκαιο και θα ακολουθήσει η τελική, η τελεσίδικη απόφαση από τα εθνικά δικαστήρια. Και υπάρχει δυνατότητα, αν δεν ε, ικανοποιηθεί, ε, να προσφύγει και στο δικαστήριο του Στρασβούργου ενδιαφερόμενος. Αυτή είναι η εικόνα, αν θέλουμε, ας πούμε, κάπως ανάγλυφα να δείξουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πώς αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που υποβάλλονται σε αυτό ενώ αυτό δεν είναι αρμόδιο. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, δέχεται πολλές ε, ε, περιπτώσεις, 61.300 πέρσι. Και τώρα ε, περιμένουν πάνω από 140.000 να εκδικαστούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύει αποτελεσματικά με τις υποθέσεις αυτές το δικαστήριο. Πόσο συχνά δέχεται καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Οι στατιστικές του 2010 δείχνουν ότι 13% των υποθέσεων που θεωρήθηκαν μη, θεωρήθηκαν παραδεκτές, δηλαδή περίπου 10% όλων των υποθέσεων απορρίπτονται διότι θεωρείται, θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Και άλλε απορρίπτονται, αλλά για άλλους λόγους θεωρούνται μη παραδεκτές, όπως δεν έχουν εξαντληθεί τα εγχώρια, ένδικα μέσα κλπ. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά αφού αφορούν υποθέσεις όπου όλες οι καταγγελίες θεωρήθηκαν μη παραδεκτές διότι ήταν εκτός αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Υπάρχουν και άλλες ε, καταγγελίες ε, που για άλλους λόγους ε, κρίθηκαν μη βαραδεκτές. Αυτές απορρίπτονται με μια συνολική φόρμουλα όπως λέμε και δεν είναι δυνατόν να τις μετρήσουμε τις υποθέσεις αυτές τελευταίες. Πάντως παρόλα αυτά μπορούμε γενικά βλέποντας την, πρακτική του δικαστηρίου μπορούμε να συναγάγουμε δύο συμπεράσματα. Πρώτον φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με τα όρια του δικαστηρίου και τις αρμοδιότητες και το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης, αλλά αυτό δεν είναι το πιο συνηθισμένο αίτιο ε, για να κρυθεί μη παραδεκτή μια υπόθεση. Εν μέρει αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αντίθεση με το χάρτη το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης δεν περιορίζεται ε, στην εφαρμογή του δικαίου συστήματος. Ένα άλλο, όταν είναι τάρτης βαθμίδας και πρέπει να κρίνει αποφάσεις ε, από τα εθνικά δικαστήρια. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Αυτό συμβαίνει συχνά και εκεί ε, πολλές απορρίπτονται ως μη παραδεκτές. Λοιπόν, ε, γενικά μπορούμε να προσθέσουμε ότι άλλα μεγάλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Και γενικά οι πολίτες και οι δικηγόροι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ε, σε αυτές τις υποθέσεις να ε, προσφύγουν ε, συχνά στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγγελίες για τις εθνικές αποφάσεις και την απονομή της δικαιοσύνης σε εθνικό επίπεδο. Και παραπονούνται εκείνοι και για το πώς εφαρμόζουν τα εθνικά δικαστήρια το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό είναι πιο συνηθισμένο. Επίσης, καλό είναι να δούμε λίγο ιστορικά την εμπειρία μέσα από το μηχανισμό της σύμβασης. Θυμάστε τη δεκαετία του 90 κάποια και κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ε, μπήκαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και προσυπέγραψαν τη σύμβαση και έτσι ε, οι πολίτες, για τους πολίτες αυτούς ε, άνοιξε νέα μέθοδος προσφύγης. Παλιά είχαν τα εθνικά δικαστήρια και καμιά φορά είχαν και τη δυνατότητα να προσφύγουν σε φορείς και σώματα των Ηνωμένων Εθνών. Και μετά που προσυπεγράφει η συνθήκη, η σύμβαση άνοιξε νέα δυνατότητα που συγκρίνεται με το, τη θέση σε ισχύ του χάρτη. Πάντα υπάρχει μία περίοδος αρκετών ετών μετά την ε, προσχώρηση όπου συσσωρεύεται γνώση για τις επακριβείς διαδικασίες, τα ωριά της, το πεδίο εφαρμογής. Δεν είναι τόσο γνωστά από την αρχή όλα αυτά. Οπότε στην αρχή είναι λιγότερες καταγγελίες και πολλές είναι μη παραδεκτές. Μετά σημειώνεται μία εξέλιξη ε, ως προς αυτό, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πάντως είναι δύσκολο να δείξουμε πούμε, σαφείς και σταθερές τάσεις σε αυτό το ζήτημα. Τι κάνει το δικαστήριο στην προσπάθειά του να αποκριθεί στην ανάγκη για σαφήνεια σχετικά με το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι δικαστικό σώμα το δικαστήριο βέβαια και το πώς αντιμετωπίζει και τις ε, προσφυγές ε, και τα αίτια που παρουσιάζει στις αποφάσεις έχουν να κάνουν με το ρόλο που έχει. Δεν μπορεί να συμβουλεύει τους ε, προσφεύγοντες. Πάντως δίνεται έμφαση από το δικαστήριο στην ενημέρωση και το Συμβουλίο της Ευρώπης κάνει πολλά και για να στηρίξει δημοσιεύσεις και τη διάδοση πληροφοριών και οργανώνει και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης δημοσιεύτηκε ένας οδηγός για, τις, να, υπάρχουν, για να είναι παραδεκτές οι υποθέσεις. Αυτό έχει να κάνει και με τα όρια αρμοδιότητας. έργα που θα αναπτυχθούν ε, είναι ένας κατάλογος παραδεκτών υποθέσεων που θα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα οδηγούνται στον κατάλληλο διάβλο μέσα από ερωτήσεις και μπορούν, θα μπορούν να φτάνουν μέχρι το Στρασβούργο να απαντήσουν ικανοποιητικά ε, σε ερωτήσεις που δείχνουν ότι μπορεί να είναι αρμόδιο αυτό το δικαστήριο. Για πολλά χρόνια, αν δούμε στο παρελθόν, στην προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρώτα χρόνια του δικαστηρίου υπήρχε μια πρακτική όπου ενημερώνονταν απευθεία οι ενδιαφερόμενοι όταν προσέφευγαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παλιότερα και στο δικαστήριο ότι μπορεί να κρυθεί μη παραδεκτή η υπόθεσή του, η καταγγελία του. Και καμιά φορά υπεδείκνυαν και άλλους αρμόδιους φορείς. Όμως, επειδή δεν έχει παραπεριορισμένους πόρους στο δικαστήριο και έχει ε, όλο ένα αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων υποθέσεων εχειριστεί, σταμάτησαν να τα κάνουν όλα αυτά. Και τώρα έχουν νέα όργανα όπως τον κατάλογο για τα παραδεκτά και τις ερωτήσεις για να κρυθεί το παραδεκτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, για την πρόληψη των βασανιστήριων, ε, επίτροπος υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι δέχονται πολλές επιστολές και απαντούν σε πρόσωπα των οποίων οι προσφυγές δεν ε, αφορούν τους φορείς στους οποίους θέλονται και τους παραπέμπουν στο σωστό φορέα. Αυτό που δεν γίνεται είναι να γίνει άμεση αναπομπή των προσφυγών που υπευλήθησαν σε ένα φορέα σε έναν άλλον εκτός και αν υπάρξει μια επιστολή που παραπέμπει στο δικαστήριο. Γιατί η άμεση μεταφορά, η μεταβίβαση, η διαβίβαση δημιουργεί προβλήματα με τους δικαστικούς φορείς. Γιατί είναι σαν να προδικάζεται το παραδεκτό. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των. Ε, προκειμένου περί τη Επιτροπή Πρόληψη Βασανιστήριων υπάρχουν ειδικού κανόνες, ειδικοί κανόνε εμπιστευτικότητα και θεωρούν ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται και να κοινοποιούνται οι επιστολές, για παράδειγμα, των φυλακισμένων σε τρίτους φορείς, οπότε δεν παραπέμπουν άμεσα. Οποιοδήποτε μηχανισμός ε, ανα, ε, διεύθυνση προς άλλες, άλλους φορείς τέτοιων προσφυγών θα πρέπει να τα λαμβάνει αυτά υπόψη αναπροσανατολισμού ας πούμε αυτών των προσφυγών. Τέλος, δύο λόγια για την αρχιτεκτονική των, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, μου φαίνεται σημαντικό όταν μιλάμε για τις δυνατότητες και τους διάφορους φορείς που είναι αρμόδιοι σε αυτό το τομέα, αν και τώρα ο στόχος πάνω απ' όλα είναι να διευκρινίσουμε την εφαρμοσιμότητα του χάρτη, αυτές οι ε, επικοινωνίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια ευρύτερη εικόνα, ούτως ώστε να κοινοποιούνται όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν και στα πλαίσια του ημεδαπού ε, δικαίου και του ενωσιακού. Έτσι θα περάσει το μήνυμα σωστά. Δεν θα περνάει δηλαδή το μήνυμα ότι δεν έχετε δικαιώματα που να απορρέουν από το χάρτη, αλλά θα υποδεικνύονται οδοί διάβλη για να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος και να βρει το δίκαιο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και βλέπω πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες ήδη να προκύπτουν όπως ας πούμε αυτός ο κατάλογος, οι ερωτήσεις για το παραδεκτό, πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά. Προχωρώ και δίνω το λόγο στον κύριο Λοτάρσκι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε που μας καλέσατε σε αυτό το εργαστήριο το τόσο ενδιαφέρον. Ε, σας ε, ε, υπενθυμίζω ότι υπάρχει δυνάμει του κανονισμού του 2001 και αρχίσαμε να λειτουργούμε το 2004 να λειτουργεί η υπηρεσία μας. Έγινε αυτός ο ορισμός από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Θητεία πενταετής 50 άτομα απασχολούν εδώ στις Βρυξέλλες. Και το βασικό, ε, βασικό βασικό σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και ιδίω όσον αυτό το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο γίνονται σε αυτά από τα θεσμικά όργανα και τι υπηρεσίε τη βεβαίω. Θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσο υπάρχει συμφωνία των δικαιωμάτων σε σχέση με τη με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, το θέμα δεν είναι τώρα το θέμα του άρθρου 16 τη Συνθήκης της Λισαβόνας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, αυτό περιέχεται και στο χάρτη τώρα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε επίσης και η αρμοδιότητά μα είναι να προστατεύουμε ε, τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Το, το οποίο ε, οδηγεί και στην ε, ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να σέβονται οι θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες. Τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε τις τρεις ευμένες δραστηριότητε για να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Πρώτα πρώτα με συμβουλές, Γίνεται αυτό μέσω τη νοθή δραστηριότητα. Δεύτερον, έχουμε και υποπτική δραστηριότητα, γιατί ακριβώ ε, εκεί ρυθμίζουμε τα των καταγγελιών. Δηλαδή, άρα, επομένω, είναι εν μέρη μόνο δραστηριότητα μα αυτέ οι καταγγελίε. Και ε, μιλούμε επίση για το τι είναι μεταξύ των δεδομένων που σε όλα τα θεσμικά όργανα και επίση παρέχουμε και τι συμβουλέ μα σε συγκεκριμένα σημεία. Ε, τώρα, για Δεν είναι επομένω η διεκπαιρέωση των καταγγελιών. Είναι μόνο ένα μέρος των εργασιών του EDPS, της υπηρεσίας μας. και έχουμε 100-120 καταγγελίες ε, ετησίως, επομένως ε, σχετικά Λίγε είναι αυτέ οι καταγγελίε σε σχέση με αυτό που ακούσαμε σήμερα, για το τι γίνεται με, με, με τι χιλιάδε των εθνικών παραπώνων, όπω εξηγήθηκε σήμερα το πρωί. Επομένω, βλέπω ότι έχουμε 100-120. Ε, ίσως έχουμε λίγο περισσότερε, ε, γιατί υπάρχει αυτή η για φέτο. Σιγά-σιγά αυξάνεται. Και τι κάνουμε όταν ε, λάβουμε αυτή την καταγγελία. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι έχουμε ε, πολύ χρόνο με προθεσμίε άνετε για τη διεκπαιρέωση. Ξεκινάει μια έρευνα, ανταλλαγή δηλαδή ε, επιστολών, ε, επαφές μπορεί να γίνουν και επιτόπου, προσβασιμότητα σε όλα τα δεδομένα που έχουν οι υπηρεσίες, ε, χωρίς περιορισμούς, είτε είναι διαβαθμισμένα, είτε είναι ιατρικά. Όχι, δεν κοίταμε βέβαια τα προσωπικά δεδομένα, αλλά πάντοτε πάμε παντού για να δούμε ακριβώ πώ γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Και κατόπιν ε, λαμβάνουμε κάποια. Και να έχει διαφορά μα σε σχέση με τον ε, διαμεσολαβητή. Ε, Εμεί δεν εκδίδουμε συστάσει, αλλά δεσμευτικέ αποφάσει. Να σταματήσει τα διεξουσία κάποιων δεδομένων. Ο διελέγκτη διατάσσει την αποκατάσταση, τη διόρθωση δεδομένων από κατάσταση κατάσταση. Επομένως, έχουμε αυτές τις 100 εκατονίξεις καταγγελίες. Έχουμε περίπου επίση και 70% ή 17% λέει ο μιλητής, των 70-70% ε, από απαράδεκτες καταγγελίες. Είναι αυτό φαίνεται πολύ. Ε, ο λόγος είναι ότι πολλές φορές είναι θέμα των ε, ιδρυτικών αρχών ή ε, έχουμε να κάνουμε με νομικό πρόσωπο. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε ή, είναι η καταγγελία κατά ε, μη κοινοτικού οργάνου. Γιατί μόνο τα κοινοτικα όργανα είναι η δική μας ομιλία. Αυτό το οποίο κάνουμε ε, δεν είναι το να τα στέλνουμε σε άλλες αρχές αμέσως. Ακριβώς όπως εξήγησαν οι προλαλήσαντες. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι το ότι Θεωρούμε ότι εάν αναπέμψουμε, διαβιβάσουμε σε άλλη αρχή ε, την καταγγελία, θα κάνουμε και εμείς παραβίαση των ε, ευαίσθητων δεδομένων. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το ότι η διαχείριση, η διεκπαιρέωση θα γίνει με τρόπο εμπιστευτικό. Και ε, ερχόμαστε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους μόνο αν είναι απαραίτητο, απολύτως πούμε, κοιτάμε αν είναι πρώτα-πρώτα παραδεκτέ οι καταγγελίε. Ε, Του λέμε γιατί είναι απαραίτητες ή αν είναι. Και αν μπορούμε, προσπαθούμε να τους πούμε δει ποιοι είναι οι αρμόδιοι και να πάνε εκεί οι παραπονούμενοι. Όλα η επιλογή πάντοτε αφήνεται ή στον ε, καταγγέλλοντα για το αν θα προσφύγει ή όχι εκεί που πρέπει. Υπάρχουν λόγοι βάσιμοι γιατί δεν θέλει ο καταγγέλων να παραπονεθεί αλλού. Πάντως, επίσης σας αναφέρω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδιαίτερη σχέση ημών και του διαμεσολαβητού. Πριν από λίγα χρόνια υπογράψαμε ένα μνημόνιο κατανόηση. Έχουν επομένω ε, κάποιε πληροφορίε ε, που είπαμε ότι θα, τις, ε, θα γίνει ανταλλαγή εάν ε, αν είναι κάτι εκείνο ενδιαφέροντο, θα υπάρχει επαφή. Αν κάτι ενδιαφέρει και εκείνου και εμά. Και έτσι προσπαθούμε να κρίνουμε κάθε φορά ποιο θα το διεκπαιριώσει. Αν είναι κακοδιοίκηση και υπάρχουν κάποια στοιχεία μόνο που έχουν σχέση με τα δεδομένα, τότε ο δημοσιολογητής θα το αναλάβει. Πάντως, γενικώ δεν διαβάζουμε υποθέσεις στους εθνικούς φορείς προστασίας δεδομένων. Πάρα πολλές λοιπόν είναι οι απαράδεκτες καταγγελίες και προσπαθούμε επομένως να ενημερώσουμε και γι' αυτό και έχουμε και μια σελίδα στο, στο site τις υπηρεσίες μας και εξηγούμε τα του παραδεκτού. Πέρσι δε είχαμε και, όπως είπε ο προλαλής σας, ή κάποιος από τους τέλο πάντων, ιδιαίτερο έντυπο. Και κατά αυτόν τον τρόπο παρέχεται ενημέρωση για το τι είναι παραδεκτό. Εντύπωση μου είναι πάντως ότι δεν τα πετύχαμε τόσο αυτά τα οποία θέλουμε. Ε, δεν μπορεί να λέω ένα mail, ε, κάποιον τον τρόπο. Ε, έχουμε ε, επιπλέον δουλειά κάθε και οπότε τους λέμε ότι θα πρέπει να απευθυνθούν σε άλλο φορέα σε έλεγχο Έτσι γίνεται όταν είναι κατάφορα παράδεκτο κάποια καταγγελία. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν τώρα δώσουμε το λόγο στην Μάργαρετ για να μας παρουσιάσει αυτή την διαδικτυακή πύλη ή Justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, σας θυμίζω ότι έχετε την θυσία μας έκθεση λάβει όσον αφορά τον χαρτί και επίσης εδώ έχετε κάποια αριθμητικά στοιχεία για τον αριθμό των επιστολών που λαμβάνουμε εκεί στη σελίδα 17 επίσης έχετε στοιχεία σε σχέση με το πώς πρωτοκολούνται οι καταγγελίες. Το πρόβλημα είναι ότι το μήνυμα αυτής της εκθέσης είναι ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης. Και αυτό ήδη το 2010 διαπιστώθηκε στον αυτή τη στρατηγική, ούτω ώστε να υλοποιήσουν το χάρτη. Και είπαμε ότι έτσι πληροφόρηση και επικοινωνία θα προσπαθήσουμε να βελτιωθεί και βλέπουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την επικοινωνία γιατί τα τελευταία χρόνια προσέξαμε ιδιαίτερα το χάρτη αλλά τώρα πρέπει να πάμε σε πιο συγκεκριμένε προσπάθειες να εξηγήσουμε περισσότερο πότε συντρέχει περί της του χάρτη και τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά που κάποιος θεωρεί ότι του έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ή στον χάρτη. Καταβάλλεται επομένω προσπάθεια από πλευρά Επιτροπή. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην επικοινωνία μα. Επίση ε, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα περίπλοκο, όπω το είπαν κάποιες φορές, σαν το πρωί, οπότε μια μεριά έχουμε τις ευξημένες προσδοκίες του κόσμου, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε νομικά θέματα τα οποία θα μπορούσε να απασχολήσουν μια εβδομάδα ένα νομικό συμπόσιο και αυτός ο συνδυασμό της υψηλή προσδοκία του κόσμου και των περιπλόκων νομικών θεμάτων οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και σε πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θέλησε να βοηθήσει συγκεκριμένα τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα θελημελιώδη δικαιώματά τους. Και ο πιο απλός τρόπος μέχρι στιγμής είναι να τους δώσουμε τον κατάλογο με τις πληροφορίες για τις ε, δυνατότητες ένδικων μέσων που έχουν στη χώρα τους. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πύλη, αυτή τη διεκτικη πυλη πύλη e-justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, ούτω ώστε να επιλύσουμε το πρόβλημα έλλειψης ε, ε, ενημέρωσης. Η Μάρκαρ θα μας παρουσιάσει αυτή τη διεκτική πύλη. Ευχαριστώ, Μανιουέλ. Καλησπέρα σας. Πολύ σύντομα θα σας ε, παρουσιάσω αυτή την ε, δικτυακή πύλη. Θα σας εξηγήσω πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανείς, πώς μπορούμε να πούμε στο, στους πολίτες, ποιοι είναι οι μηχανισμοί ε, που υπάρχουν στα κράτη-μέλη ένδικων μέσων. Εδώ και χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες στα κράτη-μέλη στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με εθνικά προγράμματα ή προγράμματα μεταξύ δύο, τριών ή τεσσάρων κρατών μελών Ο αριθμός των πολιτών που ζει εκτός του κράτους του ε, μεγαλώνει και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις. Οι στατιστικές είναι σαφείς. 11,3 εκατομμύρια άνθρωποι το 2008 ζούσαν σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό το δικό τους. Το 2008 ουσιαστικά ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε την ε, τεχνολογία για να εξορθολογήσει και να πλουστεύσει τις διαδικασίες και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη των πολιτών. Επίσης, ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την προσπάθειά μας στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ε, και να εμπλέξουμε περισσότερα όχι μόνο λίγα ε, σε αυτό που κάνουμε. Το θεσμικό πλαίσιο είναι. Το Μάιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μία ανακοίνωση με τίτλο προς μια στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικής δικαιοσύνης εν συνεχεία. Το Νοέμβριο του 2008 ακολούθησε ένα σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη το Κοινοβούλιο επίσης πλάκι στενά και υιοθέτησε ένα ψήφισμα το Δεκέμβριο του 2008 και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη ε, με οριζόντιο τρόπο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις στον τομέα της αστικής, ποινική και διοικητικής δικαιοσύνης, όπως είπε. Τέλος, δεδομένου του φιλόδοξου αυτού προγράμματος για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, στο τέλος του 2012 θα γίνει μια πρόταση για μια νομική βάση για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Οι βασικές αρχές για την προσπάθειά μας στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ότι έχουμε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση, θα δημιουργήσουμε κεντρικές βάσεις δεδομένων με στόχο να ε, συνδεθούν οι εθνικές βάσεις δεδομένων ούτως ώστε οι πληροφορίε να είναι στη διάθεση όλων. Κάνουμε μια προσπάθεια βαθμιαία. Ξεκινήσαμε με κάποιε πληροφορίε τι οποίε εμπλουτίζουμε συνέχεια. Είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα. Είναι μια διαδικασία. Και υπάρχουν 20 υποπρογράμματα από διασύνδεση ας πούμε, των κτηματολογίων, των επιχειρηματικών μητρών, των μητρών αφαιρεγγιότητας των επιχειρήσεων κτλ. κτλ. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κρατημέλη, με τα άλλα θεσμικά όργανα, με τους επαγγελματίες του κλάδου, του νομικού κλάδου, με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, προφανώς, και το περιεχόμενο στη διαδικτυακή πύλη όλο είναι σε όλες τις γλώσσες τις επίσημες εκτός από τα Ιρλανδικά. Το Ιούλιο του 2010 ξεκίνησε να λειτουργεί η πύλη σε 22 γλώσσες με 12.000 σελίδες. Το τέλος του 2011 θα έχουμε την επικυρωμένη εκδοχή και θα έχουμε και δελτία για τα δικαιώματα των θυμάτων, των κατηγορουμένων, καθώς και σελίδες και δελτία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Προσπαθούμε να πλουστεύσουμε την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των πηγών ενημέρωση. Έχουμε και άλλες ε, ιστοσελίδες της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης ε, έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικά και εμπορικά θέματα που θα ενσωματωθεί στην πύλη. Θα προσθεθούν πολλές πληροφορίες για την οδηγία καθυστερημένων πληρωμών και για άλλα στοιχεία για μικρές απαιτήσει, ε, την Ευρωπαϊκή Εντολή για τις πληρωμές κτλ. Το 2012 Αυτά θα είναι τα βασικά κεφάλαια, ε, πηγές δικαίου, ε, δικαστικά συστήματα, ε, ένα τμήμα για τα δικαιώματα, επίλυση διαφορών κτλ. Έχουμε κάποιες σελίδες που τις διαχείριζεται η Κομισιόν και έχουμε και σελίδες των κρατών μελών που τα κράτη-μέλη είναι ιδιοκτήτε και κάνουν την επικαιροποίηση στη γλώσσα του και εμεί τα μεταφράζουμε. Και αυτό το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά. Επίση, θα έχουμε και εργαλειοθήκε, πρακτικέ. Αν θέλει, Φερρυπίν, να βρει, α πούμε, τη Γαλλία και θε να βρει έναν δικηγόρο στη Γαλλία, ο οποίο μιλάει Ισπανικά και εξειδικεύεται στο οικογενειακό δίκαιο, θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο στην πύλη για να δεις Πού μπορεί να βρει αυτό το δικηγόρο και τα στοιχεία του βέβαια. Η σελίδα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πύλη ε, είναι στο τμήμα τα δικαιώματά σου. Είναι σε αυτό το τμήμα της πύλη, Παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι ξεκινάει. Και έχουμε μια ε, σελίδα εισαγωγική με όλες τις βασικές πληροφορίε για τους φορείς που εμπλέκονται, να, ε, σε ποιο να απευθυνθείς, με ποιο να σε και πότε ε, ισχύει ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τι εθνικέ σελίδε για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, καλύπτουν τα εθνικά δικαστήρια, του εθνικού θεσμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του ε, ombudsman, εξειδικευμένου φορεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οποιασδήποτε άλλε πληροφορίες θέλουν να δώσουν τα κράτη-μέλη πέρα από του διαμεσολαβητέ και όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Αυτή είναι η αρχική σελίδα της πύλης υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Μπορείς να προσωποποιήσεις την πρόσβασή σου, να δεις τι προτιμήσεις έχεις γλωσσικές ε, και μπορείς επίσης να ζητήσεις και την επικαιροποίηση όταν γίνεται να σου έρχεται. Αν καταχωρηθείς και ζητήσεις ενημέρωση, θα πάρεις μια κοινοποίηση στο email σου, ούτως ώστε οποτεδήποτε κράτη-μέλη ενημερώνουν τη σελίδα τους για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το μαθαίνεις μέσω του email σου. Ε, οι δυνατότητες αναζήτησης επίσης βελτιώνονται συνέχεια. Αυτή η εκδοχή θα είναι στο διαδίκτυο το Νοέμβριο του 2011. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός, μιας σελίδας ενός κράτους μέλους πώς μπορείς να βρεις ένα διαμεσολαβητή στην Ισπανία. Και εδώ βλέπετε όλες τις σελίδες των υπόλοιπων κρατών μελών. Ένα άλλο παράδειγμα μιας γαλλικής σελίδας α, στα αγγλικά γαλλικής νομολογίας δηλαδή στα αγγλικά Τώρα, για την χρήση της πύλης. Έχουμε μέχρι 50.000 επισκέπτες το μήνα, 35.000 το Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε. Το, η πύλη αυτή δεν έχει προωθηθεί από την ημέρα που ξεκίνησε πολύ, δεν έχει διαφημιστεί πολύ και η χρήση εξαρτάται πολύ από το πώς τα Υπουργεία Δικαιοσύνης των κρατών μελών την προωθούν. Στη Ρουμανία, ε, σε κάθε σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχει ένα link για αυτή την ε, ε, δικτυακή πύλη. Γι' αυτό το 25% των επισκεπτών είναι Ρουμάνοι. Έτσι εξηγείται αυτό το γεγονό. Δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία αν δεν τα προωθούμε. Γι' αυτό φέτο θα επιταχύνουμε τι προσπάθειέ μα και εμεί, αλλά και το 2012, Κομισιόν και κράτη-μέλη, ούτω ώστε να στοχεύσουμε την προώθηση. Όταν ετοιμάσουμε αυτές αυτά τα δελτία για τα δικαιώματα των θυμάτων, ε, των κατηγορουμένων κτλ τα fact sheet, δηλαδή τα δελτία που σας ανέφερα προηγουμένως. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται και δουλεύει στον τομέα, θα θέλαμε να μας βοηθήσει. Ε, θέλουμε να σας δώσουμε, παραδείγματος χάρη, ε, σήματα, να τα βάλετε στις ε, ιστοσελίδες σας, για να υπάρχει ένα link με το πόρταλ αυτό. Ε, θα γίνει μια γενική εκστρατεία το 2012 μέσω των νομικών σχολών, ε, μέσω, και γραφείων κτλ. για να προωθήσουμε την ε, πύλη αυτή. Τα Υπουργεία Δικαιοσύνη των κρατών μελών φυσικά εμπλέκονται πολύ σε αυτό που κάνουμε και έχουν τουλάχιστον ένα link στην ιστοσελίδα τους όλα τα Υπουργεία. Αν θέλετε λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί μας ή να επισκεφτείτε την πύλη. Μην αμελήσετε να το κάνετε. Θα ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε τις απόψεις σας για τις σελίδες μας ε, και οποιασδήποτε προσπάθειες κάνετε για να την προωθήσετε είναι ευπρόσδεκτη. Η προσθέμενη αξία είναι ότι ε, δημοσιεύονται σε όλες τις ε, γλώσσες, τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προσπελάσιμα βέβαια από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Μάργαρετ. Θα δώσω το λόγο τώρα στο κοινό. Δεν ξέρω ποιο θα... ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ανακουφίστηκα λίγο, γιατί ήμουν μόνη εδώ βουλευτής να εκπροσωπώ 500 εκατομμύρια. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Τώρα όμως ε, ήρθε κι άλλος. Δύο ερωτήσεις. Μία στον David Lowe να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ε, υπάρχουν, να πούμε ότι υπάρχουν εμπόδια από την Κομισιόν. Να είναι καθαρό ότι η Κομισιόν, για να το πούμε ήπια, είναι απρόθυμη να ασχοληθεί καν. Ακόμα και όταν είναι σαφές ότι πρέπει να το κάνει. Και πρέπει να τονίσουμε ότι ένα εμπόδιο που έχουμε στην Επιτροπή, έχουμε πολλά, αλλά ένα πραγματικό εμπόδιο είναι αυτό, ότι η Κομισιόν δρά, λες και είναι δικαστήριο. Ενώ υπάρχουν δύο διαφορετικοί φορείς. Άλλο το δικαστήριο. Δεν πρέπει εκείνη να το κάνει αυτό. Πρέπει να διευκολύνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έτσι προβλέπουν οι συνθήκες. Κάτι άλλο που βλέπουμε συχνά. Η πρόσβαση στα έγγραφα από γονείς κλπ. Και εκεί Δημιουργεί κάποια μηχανία το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν το προχωρεί το πράγμα και δεν ακούει τι της λέει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και κοιτάει να αποφύγει να ασχοληθεί με αυτό το θεμελιώδες δικαιώματα που είναι και στο χάρτη και πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στις διοικήσεις και παντού. Έχουμε λοιπόν και εμείς αυτές τις δυσκολίες και δεν φαίνεται η παρουσία μας ε, στους πολίτες και στις σκανδιναβικές χώρες δεν ε, τα ξέρουν γιατί δεν έχει ε, μεταφραστεί και το όνομα της Επιτροπής. Και δεν ξέρουν δηλαδή τι, ποια είναι η Επιτροπή, τι κάνει και πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Τώρα, το βασικό μου ερώτημα αφορά το δικαστήριο. Γιατί νομίζω και συμφωνούμε απόλυτα και αναφέρομαι σε αυτά που είπαμε στην πρωινή συνεδρία ότι τα ατομικά δικαιώματα θα πρέπει να τα καταπιάνονται σε εθνικό επίπεδο. Αν υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να την ακολουθούν την απόφαση αυτή και τα εθνικά δικαστήρια. Εγώ έχω υποθέσεις από τη Δανία και ξέρω και άλλες από άλλες χώρες γιατί δεν, έρχονται, δεν έρχεστε σε επαφή με τα δικαστήρια ούτως ώστε η προδικαστική απόφαση που θα λάβει το Εθνικό Δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη την ενωσιακή νομοθεσία, το δίκαιο της Ένωσης. Στη χώρα τη δική μου, τα δικαστήρια δεν ε, θέλουν να ρωτήσουν και να ενημερωθούν από πριν. Ίσως επειδή θεωρούν ότι ένα δικαστήριο δεν πρέπει να ρωτάει, να απαντάει μόνο πρέπει. Ε, είναι ενάντια στη φύση τους θεωρούν. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Κομισιόν δεν ενδιαφέρονται όμως. Άρα, μπαίνει ένας φαύλος κύκλος και όλοι πάνε στο Στρασβούργο, θέλουν να πάνε στο Στρασβούργο, με όλο το σεβασμό και εγώ ήμουν ε, χρόνια και στην Επιτροπή τη Νομική, αλλά Ε, αυτά είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί κάποιον να τον στείλει στο Στρασβούργο γιατί θα χαθεί. Επανέρχονται λοιπόν και μας ρωτούν πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε εθνικό επίπεδο. Εκεί τι, πώς να κατευθυνθούμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν υπόψη τα η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει ερωτήματα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με, ε, στα εθνικά δικαστήρια. Αυτό ίσως θα ανταποκρινόταν περισσότερο προς, την, το ρόλο τους όπως τον ε, αντιλαμβάνονται. Ευχαριστώ. Είναι καλό που έχουμε τους εκπροσώπους των δύο δικαστηρίων εδώ μαζί, γιατί θα δούμε τι θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα ε, με τις ε, κρεμμύς υποθέσεις. Είπατε ότι υπάρχει, υπάρχουν χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να ξεριζωθούν τα προβλήματα μετά την προσχώρηση, μέχρι να, γίνουν κατανοητό, να γίνει κατανοητό ποιε είναι παραδεκτές κλπ. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι 38% όλων των υποθέσεων αφορούν Ρωσία και Τουρκία και γι' αυτό δημιουργείται συμφόρηση στη, στα δικαστήρια. Περνώ έτσι στην επικουρικότητα και στην ανάγκη οι προσφορούσες χώρες να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα, τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση να ενσωματωθούν στην ημεταπή νομοθεσία. Ε, όλα τα ενωσιακά όργανα θα πρέπει όταν επικυρωθεί η σύμβαση να την τηρούν και θα μην μειωθεί η ανάγκη προσφυγής στο Στρασβούργο. Ε, με την επικουρικότητα θα φροντίσουμε με όπως η υπόθεση ΕΝΕΣ να μην πάει στο Στρασβούργο και να ε, γίνει ε, χειρισμός σε ενωσιακό επίπεδο. Μπορεί να παρακαμφθεί το δικαστήριο αν ένας ε, κάποιος προσφύγει ας πούμε κατά του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα και τότε η υπόθεση θα πάει στο ε, δικαστήριο του Στρασβούργου. Οι θεσμοί της Ένωσης θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουν ότι η, η ε, νομολογία του δικαστηρίου να τηρείται. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ε, φροντίζομαι η νομολογία να λαμβάνεται υπόψη γιατί αν συμβεί αυτό θα μειωθεί και το μποτιλιάρισμα που συμβαίνει στα ε, δικαστήρια. Ευχαριστώ, πολύ, λέει ο κ. Μποσινάρου. Η ερώτησή μου κάπω είναι στο μήκο σχήματο των όσων λέγαμε το πρωί γιατί είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε εδώ πέρα τον εκπρόσωπο ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων διότι προκύπτει σαφώ ότι εις κάποιες ε, πάρα πολύ βασικές ε, υποθέσεις όπως η παραβίαση των, ε, των του δικαιώματος εις την προσβασιμότητα στα ελεύθερα ΜΜΕ δεν θα αποτρέχει ποιε χώρε, χώρες αλλά πρόσφατα υπήρχε πρόβλημα σε δύο, τρεις, τέσσερις χώρες Επομένω, θα πρέπει να δούμε πώς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε εμεί με εσά και με το Συμβούλιο της Ευρώπης διότι έχουμε Αυτά τα οποία έχει αξιολογήσει ο, ο, ο αρμόδιος τέλο πάντων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ελεγκτής και, και, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με, την, ε, και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, στα κράτη-μέλη, για θυμάμαι τι είπαν για το ε, τι τύπο για ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη νομοθεσία και θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίφημη υπόθεση Handicide που έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντική υπόθεση για το εδώ για των δικαιωμάτων και επίσης υπάρχει και θέμα κριτηρίων της Κοπενχάγης όπως το το πρωί και έχει σχέση με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες χώρες οπότε τώρα τα κράτη-μέλη όμως δεν τους ζητείτε να υλοποιήσουν τα στάνταρ για, ας πούμε, για την ελευθερία των ΜΜΕ ακριβώς όπως με τα κριτήρια τα οποία ε, θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό διότι η Ευρώπη ε, λέει ότι είναι πρωταθλητές στα θρονοδιώματα μα και έχουμε από την άλλη μεριά Κίνα και Ρωσία που τους κατηγορούμε ότι δεν εφαρμόζουν δικαιώματα για τα μη Όμως εδώ μέσα στο σπίτι μας έχουμε ξεκάθαρες κατάφορες περιπτώσεις παραβίασης αυτών των κριτηρίων. Και δεν κάνουμε τίποτα. Εσείς τι λέτε. Your evaluation to be somehow... Παρακαλώ, επομένω. Πώς θα αξιολογείτε τα πράγματα. Πώς μπορούμε να έχουμε κάποιο ρύθμιση δεσμευτική. Για καθημερινή χρήση, όχι για πολιτικές εξαγγελίες. Γιατί με προβληματίζει πάρα πολύ το θέμα. Καλά, υπήρχαν θέματα πριν την ε, προσχώρηση. Μετά την προσχώρηση, τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι επικουρικότητα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει κανείς τότε. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Γιατί μπαίνει η ερώτηση. Στην παρουσίαση μου δεν είχα πολύ χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες. Ένα θέμα που έχουμε αντιμετωπίσει ως Εθνικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά κάτι που αφορά και άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αν θα πρέπει ε, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να τις αλλάξουμε, ούτως ώστε να επιτραπεί κάποια δράση. Αν δεν είσαι διάδικος σε εθνικές διαδικασίες, ούτως ώστε ε, να δεις τι θα γίνει σε σχέση με αυτήν την αντίφαση. Από τη μία δεν είσαι διάδικος, αλλά από την άλλη στο δικαστήριο του Στρασβούργου μπορείς να πας ως διάδικος. Η χάρτα τώρα είναι δεσμευτική και το, η νομολογία του δικαστηρίου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρχίζουν να έχουν όλο και πιο παραπλήσια νομολογία. Ποια είναι η άποψή σας ε, μίλησα με τον επικεφαλής του Μητρώου την περασμένη εβδομάδα, γνωρίζει αυτά τα θέματα και αν προταθούν κάποιες αλλαγές, το δικαστήριο θα πρέπει να τις κάνει αυτές τις προτάσεις. Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, πρέπει να τις κάνει το δικαστήριο τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές, να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις για την επικοινωνία. Έχετε κάνει κάποιες αναλύσεις ή κάποιες αξιολογήσεις ε, για το τι είναι πιο αποτελεσματικό. Είναι ένα site στο ίντερνετ. Είναι κάποιες απαντήσεις ε, πιο λεπτομερείς, πιο προσεκτικές, ε, υπομορφή επιστολών για να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν υπάρχει δικαιοδοσία. Χρησιμοποιείτε κάποιες στρατηγικές επικοινωνίες συγκεκριμένες. Κάντε κάτι τέλος πάντων. Και κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσουμε τους πολίτες. Εγώ ως υπάλληλο στην Επιτροπή λαμβάνω ε, επιστολές από τους πολίτες ε, και βλέπω εκεί συμπεριλαμβάνουν ας πούμε τμήμα των απαντήσεών σας που είναι έτοιμες απαντήσεις οι δικές σας ή του Ευρωπαίου Επόπτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Προστασίας των Δεδομένων κτλ και δεν τους ικανοποιεί αυτό τους πολίτες. Επίσης, υπάρχουν ε, πολλές επιστολές από την ΑΒ χώρα. Τι σημαίνει αυτό. Φυσικά δεν πρέπει να βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, αλλά κάτι σημαίνει αυτό. Έγιναν κάποιες μελέτες, τέλος πάντων, για τις προσδοκίες που εκφράζονται μέσω των επιστολών των πολιτών. Ζητήσατε να γίνουν και ονειολογικές μελέτες για το τι σημαίνει αυτό. Ο Ντέιβιντ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για την ε, Μάργαρετ για ένα πολύ λεπτό θέμα για τις διαθεσμικές σχέσεις. Θα δώσω μια πιο μακροσκελή απάντηση για να συμπεριλάβω και άλλα θέματα, ώστε να σας απαντήσω καλύτερα. Αυτά που άκουσα από τους ομιλητές εδώ από το πάνελ Και από αυτά που άκουσα και το πρωί και από τις δηλώσεις και από τις ερωτήσεις, ε, νομίζω ότι τελικά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που προσεγγίζουμε τη διαδικασία των αναφορών στο Κοινοβούλιο, με ένα θετικό τρόπο. Λέμε στους πολίτες, εδώ είναι το Κοινοβούλιο, το καθήκον είναι να υπηρετήσει τους ανθρώπους που το εξέλιξαν. Έχουμε ένα, μια θετική αρχική στάση τουλάχιστον για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών θεωρούμε ότι καταρχάν έχουν δίκιο οι, καταρχήν έχουν δίκιο οι αναφέροντες. Δεν κάνουμε όπως είπαν, υπενήχθηκαν ή το είπαν και ρητά ε, οι υπόλοιποι ομιλητέ. Εμεί δεν περιοριζόμαστε σε αυστηρά νομικίστικες ή νομικές δικαιολογίε για το τι πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση που θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Η αναφερόμενοι απευθύνονται κατευθείαν σε εμά στο Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να περάσουν από κάποιον Ευρωβουλευτή, δεν χρειάζεται να περάσουν από κάποιο εθνικό προηγούμενο βήμα ε, ή να έχουν εξαντλήσει άλλα μέτρα. Τίποτα. Πηγαίνουν κατευθείαν, στρέφονται κατευθείαν προ εμά και του ε, απαντάμε. Μπορεί να μην του αρέσει η απάντηση, τουλάχιστον όμω σε κάθε περίπτωση απαντάμε. Δεν χτυπάνε τη λάθο πόρτα δηλαδή για θέματα, για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι προσδοκίες για το τι μπορεί να πετύχει το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την εξαίρεση λύσης για ανθρώπινα δικαιώματα είναι τελείως διαφορετικό, ε, οι προσδοκίες τελείως διαφορετικές από τις προσδοκίες που έχει από ένα δικαστήριο. Επομένως πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Και για να επανέλθω σε αυτά που είπε η Μάργαρετ για, για τα εμπόδια, για τους φραγμούς που αντιμετωπίζουμε. Ένας από τους φραγμούς είναι ακριβώ αυτός. Επειδή οι ευρωβουλευτέ είναι πιο ανοιχτοί εκφύσεω και αισθάνονται μια ευθύνη, θέλουν να δώσουν απαντήσει στους πολίτες, εμείς εξετάζουμε έναν τρόπο έτσι ανοιχτό και σφαιρικό τα θέματα στις αναφορές μας ε, και αναφορές που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φυσικά μας βάζει εμπόδια η Κομισιόν και μας απογοητεύει αυτό. Όταν αντιμετωπίζουμε θέματα που εμεί τα θεωρούμε θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, καλό θα ήταν να ακούσουμε τους, την εμπειρία των, την άμεση εμπειρία των πολιτών. Είναι απογοητευτικό λοιπόν όταν η Επιτροπή λέει ότι αυτό δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα, δεν μπορώ να ασχοληθώ ε, με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία γιατί αυτό δεν είναι ε, το σύστημα ας πούμε της ιδιοκτησίας δεν είναι ενωσιακή αρμοδιότητα. Εδώ μιλάμε για τα δικαιώματα. Μιλάμε για το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Μιλάμε για το σεβασμό της ακαιρεότητας των ανθρώπων ως πολίτες ή κατοίκου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ετούντες άσυλο. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω εκ μέρους των Ευρωβουλευτών, οι ευρωβουλευτές ε, αισθάνονται ότι τους περιορίζει η Κομισιόν στην ερμηνεία της για τις αρμοδιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη δικαιοδοσία που έχει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτό δημιουργεί κάποια απογοήτευση στην Επιτροπή Αναφορών. Άκουσα το σχεδιασμό του, της δικτυακής πύλης που έχει η Κομισιόν. Μακάρι να είχαμε και εμείς το ίδιο. Το προσπαθούμε. Ε, πόρα απέχουμε βέβαια. Και θα προσθεθεί στην πληθώρα αυτών των πυλών που υπάρχει. Και το θέμα είναι πόσοι πολίτε τελικά θα πάρουν απάντηση βέβαια. Ε, υπάρχει και, το, και η πύλη του διαμεσουλαβητή. Είναι μοντέλο για όλους μας. Βάλτε και την Επιτροπή Αναφορών, θα έλεγα εγώ, στην ε, δικτυακή σα πύλη, Ω ακόμα μία πηγή. Αλλά να ξεκαθαρίσετε απλώς ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Αυτό που έχουμε είναι αυτό το φυλάδιο, το newsletter, ε, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει συνδρομητής. Ε, που ονομάζεται το μικρό εφημεριδάκι στα γαλλικά, λεπτή Journal. Δεν τόσο τέλειο όσο μία πύλη. Είμαστε και στο Facebook και στο Twitter. Υπάρχει μια συνεχής έτσι, ενημέρωση. Α, ανανεώνται οι φίλοι μας, παρακολουθούν τη δουλειά μας. Ε, μπορείτε να δείτε τι δραστηριότητες προωθούμε. Ε, αλληλεπιδρούμε με πολύ ανεπίσημο τρόπο με τους πολίτες, ούτως ώστε να συζητάμε μαζί τους για τα δικαιώματά τους, τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να τους βοηθήσουμε. Απατώντα λοιπόν ε, στο ερώτημα της Μάρκετ, παρέκλεινα λίγο βέβαια, αλλά το βασικό θέμα είναι η επικοινωνία με τους πολίτες. Ο διάλογος μαζί τους είναι σημαντικός για το Κοινοβούλιο. Σεβαζόμαστε τα δικαιώματα και τις ε, αρμοδιότητες του δικαστηρίου, είτε είναι το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, είτε το δικαστήριο στο Στρασβούργο. Ξέρουμε πόσο δύσκολο και δαπανηρό είναι ένα πολίτη να φτάσει σε αυτά τα δικαστήρια και να καταλάβει και τι προδικαστικέ αποφάσει που εκδίδονται, γιατί δεν έχουν καμία σχέση, αισθάνονται πως δεν έχουν καμία σχέση με αυτού. Σω πρέπει να κάνετε και μια προσπάθεια να εκφραστείτε με πιο απλό τρόπο προ του πολίτε, να του εξηγήσετε ποιε είναι οι επιπτώσει μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ούτως ώστε να στρέφονται οι άνθρωποι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για απάντηση. Και να υπάρχει μια καλύτερη σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και τους πολίτες και μεταξύ όλων των υπολείπων φορέων που εκπροσωπούνται εδώ και των πολιτών. do you want to, to reply? Θα απαντήσετε. Εκτός μικροφόνου. Αυτό η ερώτηση ποια ήταν, τι γίνεται όταν τα εθνικά δικαστήρια δεν παραπέμπουν ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προδικαστικό ερώτημα. Τότε το, θέμα είναι ακριβώς ποια είναι η σχέση μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Δικαστήριου στη διαδικασία των προδικαστικών ερωτημάτων. Τότε το θέμα είναι, ε, ο κανόνας είναι, η απάντηση είναι συνεργασία ίσον. Δεν κατησχεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με τα ανώτερα, ανώτατα ελληνικά, ε, εθνικά δικαστήρια. Και επομένως με τίποτα το δικαστήριο δεν μπορεί να να υπερβεί την αρμοδιότητά του και αυτό είναι γενικός κανόνας. Φυσικά τα δικαστήρια αποφασίζουν όταν κάποιος προσφύγει εντός της ομοιότητάς τους, την οποία δεν υπερβαίνουν. Όμως, δεν γίνονται εισαγγελική αρχή τα δικαστήρια. Δεν ασκούν κανένα τους ποινική δίωξη. Αυτό τα κάνουν οι εισαγγελείς. Τώρα, τι να σου πω, μπάσκες στη ΣΥΠΑ γίνεται αλλιώς, γιατί έχουν άλλο σύστημα. Όμως, Υπάρχει πιθανότητα εάν κάποιος δεν συμφωνεί με κάποια απόφαση κάποιας πολιτείας της ΣΥΠΑ μπορεί να προσφύγει στο του Δικαστήριο 5.000 τέτοιες υποθέσεις δικάζει το Νότατο Δικαστήριο της ΣΥΠΑ και έχουν την κριτική ευκαιρία να επιλέξουν ποιε θα κρίνουν και διαλέγουν καμιά εκατοστή ετησίω. Όμως είναι διαφορετικό το σύστημα σε σχέση με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όπως έχει το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο και να αναλάβει την πρωτοβουλία που υπονοείται. Ευχαριστούμε. Για να συνεχίσουμε τώρα το ίδιο θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα σε σχέση με το πώς μπορεί να λησμονώνονται δύο δικαστήρια ακριβώ από αυτό το θέμα, διότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει κρίνει επανειλημμένα, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα των υποθέσεων, στις οποίες υποθέσεις έχει κρίνει ότι είναι αυθαίρετη η άρνηση του Εθνικού Δικαστηρίου να αναπέμψει για προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ μία υπόθεση και ίσως λέει ότι αυτό είναι και άρνηση του δικαιώματος στην δίκαιη δίκη. Είναι λέει, είναι λέει αυτό παραδιαστροπή δικαιωμάτων, λέει το ΔΕΚ complementarity. Uh, on, the questions which... Uh, τώρα, Ναι, γιατί εννοώ για την τώρα, όσον αφορά τις άλλες ερωτήσει που εν μέρη με αφορούσαν, βεβαίως και ευχαριστώ για την έμφαση που δώσατε ή στην επικουρικότητα. Έχουμε και τη διακυβερνητική διάσκεψη και Έχουμε κάποια μέτρα ούτως ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η διαδικασία, να απλουστευτεί, να είναι πιο αποτελεσματική και επίσης έχουμε και κάποια άλλα σημάδια, μηνύματα προ τα κράτη-μέλη όσον αφορά το καθήκον τους λόγω τη αρχή τη επικουρικότητα ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτα και κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Να, Πώς μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική προστασία. Και να πώς η ύλη του δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού μικραίνει. Να το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε ισχυρό. Προς τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να κάνουν περισσότερα στις εθνικές αρχές. Να, τι θέλει το δικαστήριο. η τώρα των αποφάσεων, όπως ξέρετε είναι θέμα της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και η διακυβερνητική διάσκεψη πάντως αναγνωρίζει ότι επιδέχεται πολύ βελτίωση στο σύστημα. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να επηρεάσει, να πιέσει τους Υπουργούς του Βουλίου της Και αυτό θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη εκτέλεση των αποφάσεων. Διότι ευρέως αναγνωρίζετε ότι όπως έχει σήμερα το σύστημα της εκτέλεσης των αποφάσεων δεν λειτουργεί πολύ καλά. Με τη σχέση των δικαστηρίων. Το σχέδιο κειμένου για την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, σύμβαση είναι λόγο, εκεί ορίζεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόσουν το κοινότικο δίκαιο χωρίς να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα μετά την ε, οριστική τους απόφαση εάν κάποιος προσφύγει στο Στρασβούργο έχει λεχθεί, έχει προβλεφθεί, έχει οριστεί ότι ανοίγει νέα διαδικασία και αναζητείται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα να μην είναι το πρώτο σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αυτονομία Δικαιωμάτων για να κρίνει αυτά τα θέματα. Τώρα κάθισαμε και αναλύσαμε τα, τις κατηγορίες των καταγγελιών και μελετάμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχουμε βασικά εδώ πέρα δύο τομείς, δύο κατηγορίες. Πρώτα πρώτα κάποιες, κάποια παράπονα, παραβίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε αναλύσει τις υποθέσεις αυτές και όποτε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαρθρωτικό πρόβλημα σε κράτος μέλο λόγω πολλών υποθέσεων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τη διαδικασία του, του, του, του, την πιλωτική. Και έτσι να έχουμε μια βασική απόφαση Οπότε δίνουμε κατευθυντήρες γραμμές στις εθνικές αρχές για το τι θα πρέπει καταρχήν να γίνει. Για να μην έχουμε παρόμοιες καταγγελίες και παραβιάσεις. Να, μία ανάλυση που έχουμε επαγγελμένα. Και για να φτάσουμε λέμε πιλωτικές ε, αποφάσεις. Επίσης έχουμε κάποιες αποφάσεις περί το παραδέκτου. Έχουμε κάποιες καταγγελίες που είναι παράδεκτες. Έχω εδώ πέρα μία μελέτη και αναφέρεται εκεί ποιες περιπτώσεις εκρίθησαν ε, απαράδεκτες. Για παράδειγμα, ε, είχαμε εδώ μία ενδιαφέρουσα υπόθεση που αναφέρει το πόσες είναι αυτές οι υποθέσεις επαράδεκτες. Και είπαμε ότι μόνο στην τελευταία φάση της διαδικασίας χρειάζεται να παρίστανται, να παρίσταται συνήγορος. Στις, ε, στις αρχικές φάσεις δεν χρειάζεται δικηγόρος. Και το 2010 δεν έχουμε τίποτα χαρακτηριστικά αποτελέσματα, δεν μας λένε τίποτα αποτελέσματα γιατί έχουμε κάποιες χώρες που πάει δικηγόρος αλλά έχουμε πολλές, ε, πολλά παράδεκτα και τέλος πάντων και το αντίστροφο. Και προς το δικηγόρο λοιπόν έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις παράδειγμα. Άρα δεν μπορέσαμε να μπορέσουμε να δούμε τι συμβαίνει. 20-25% γενικά απορρίπτονται από αυτές τις υποθέσεις. Ένα συμπέρασμα από την ανάλυση είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνονται και οι νομικοί και, και ο κόσμος όσον αφορά τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου και τα όρια αυτών. Merci beaucoup. Sorry. Very briefly about the, the question of Mr. Chairman about our strategies uh, of communication and what... Να σας πω για στρατηγική επικοινωνία μας με δύο λόγια μόνο. Κοιτάξτε, όποτε καθόμαστε να αξιολογήσουμε τις καταγγελίες, από προέρχονται, τι θέμα έχουν, και όποτε έχουμε επίσης ε, γενικά απαράδεκτες ε, αποφάσεις. Να έχουμε και αυτή την ετήσια έκθεσή μας που τα συζητεί. Και έχουμε εδώ και αριθμητικά στοιχεία. Οπότε κατόπιν τη αναλύση προσπαθούμε κάπω να προσαρμόσουμε την επικοινωνία μα πριν μερικού μήνε. Είχαμε πάρα πολλέ απαράδεκτε υποθέσει σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια, αυτό είναι ιδιωτική δραστηριότητα, δεν σα αφορά. Οπότε, πάντως εμείς ε, είπαμε ότι μην παραπονιέστε σε εμά για τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά θα πρέπει να πάτε σε κάποια εθνική αρχή. Αυτά κάναμε κατόπιν της έρευνας αυτή την ανάλυση. Πρόεδρος, Εκτό μικροφώνου. Merci beaucoup. Je propose de, clôturer ce... Να κλείσει αυτό το πάνελ. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο πάνελ που είναι και τελευταίο. Πρέπει να τελειώσουμε οπωσδήποτε στις 5. Ευχαριστώ για το τελευταίο αυτό πάνελ ε, που θα ξεκινήσει τώρα, που έχει σαφή στόχο. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε και παρουσιάσαμε την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο. Το απόγευμα προσπαθήσαμε να δούμε τις ε, πρακτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο πάνελ θα μας μιλήσει για το αν μπορεί να υπάρξει περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και του εθνικού επίπεδου. Αυτό το θέμα υπήρχε στην ετήσια έκθεση που ασχολείται με την εφαρμογή του χάρτη, όπου προσπάθησαμε να σκεφτούμε αν μπορούμε να βρούμε νέες μεθόδους συνεργασίας. Αν γίνεται, Φερρυπίν, να αναπέμψουμε κάποιες καταγγελίες το συζητήσαμε στο προηγούμενο πάνελ λιγάκι. Νομίζω ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να διερευνήσουμε, να σκεφτούμε τον τρόπο βελτίωσης της συνεργασίας των αρχών. Σήμερα το πρωί καταλάβουμε πούμε, ότι στο Βέλγιο γίνονται σοβαρές προσπάθειες για το συντονισμό της χώρας. Και φαντάζομαι ότι αυτή η προσπάθεια συνεργασίας μπορεί να γίνει μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επίπεδου. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε αυτές τις δυνατότητες συνεργασίας και να καταλάβουμε καλύτερα τι υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Ε, θα ακούσουμε το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στη Σόνια Μαζίνη, που είναι αντιπρόεδρος της ε, Περιφερειακής Επαρχίας Ε, του Ρέτζο Εμίλια και πρώτη αντιπρόεδρος τη Επιτροπής Ιθαγένεια Δικυβέρνησης ασμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων τη Επιτροπής των Περιφερειών. Σήμερα το πρωί ο Ντομινίκ Πουντής είπε ότι υπάρχουν 600 κέντρα όπου μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτη ε, για να φτάσει στον διαμεσολαβητή. Βλέπετε το περιφερειακό επίπεδο που μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να αποκτήσουν σάρκα και οστά τα δικαιώματα αυτά. Ε, η Σόνια Μαζίνη. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, καλό απόγευμα. Θα μιλήσω Ιταλικά, που είναι η μητρική μου. Εκπροσωπώ την Επιτροπή των Περιφαριών, που θέλει να δώσει ένα σημαντικό ρόλο στις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, και το ρόλο που μπορούν να παίξουν για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, προσπαθεί να δώσει προσανατολισμού στους πολίτες για να βρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή των Περιφερειών τόνισε σε διάφορες νομοδοτήσεις ότι παρότι η Ευρώπη έχει ένα νομικό πλαίσιο πολύ καλά διαρθρωμένο σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, στην πράξη υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε ό,τι αφορά τις εγγυήσει και την προστασία αυτών των ε, δικαιωμάτων. Επομένως, η Επιτροπή μας συμφωνεί με την Κομισιόν, όπως ε, εκφράστηκε η άποψη της, ε, από την έκθεση του 2010 για την εφαρμογή του χάρτη της ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που λέει ότι θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εντυπωσιακό που παρότι αναγνωρίζουμε αυτή την ανάγκη, δεν ε, αναφέρεται ο ρόλο ο σημαντικό που μπορούν να παίξουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές. Υπενθυμίσαμε πολλές φορές ότι με βάση το άρθρο 51 παράγραφος 1 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και από τα κράτη-μέλη όταν αυτά ενεργοποιούν το ενωσιακό δίκαιο και των συμματών στην εθνική νομοθεσία. Τα κράτη για να ενεργοποιήσουν τους κανόνες που είναι ευρωπαϊκής προέλευσης με, δρούν με βάση τους δικούς εσωτερικούς κανόνες ε, και λαμβάνουν υπόψη τις νομοθετικές και διοικητικές ε, αρμοδιότητες που υπάρχουν στα διάφορα ε, επίπεδα διακυβέρνησης. Σε πολλά κράτη-μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν νομοθετικές και διοικητικές αρμοδιότητες και σε τομείς όπου οι, οι επιπτώσεις του νοσιακού δικαίου είναι πολύ σημαντικές. Συχνά, λοιπόν, οι αρχές αυτές ε, ουσιαστικά ε, πρέπει να δράσουμε τρόπο που να σέβονται τα, τα δικαιώματα του χάρτη. Στην Ιταλία το άρθρο 117 αναγνωρίζει ε, νομοθετικές αρμοδιότητες στις περιφέρειες για την προστασία της εργασίας, της υγείας, εκεί όπου οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι πολύ σημαντικές. Στις ορισμένες ε, α, περιφέρειες Ιταλίας γίνεται σε πολλά κείμενα ε, αναφορά στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ε, περιφερειακή νομοθεσία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως την ε, διοικητική ε, αυτονομία των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μπορεί να μπουν θέματα που αφορούν την εξασφάλιση και την προστασία αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, ζητώ συγγνώμη που μιλάω πολύ γρήγορα. Το κάνω για να περιορίσω το χρόνο που μιλάω. Μην ξεχνάτε την πολιτική των ενοικίων, ε, το δικαίωμα στο απαραβίαστο της προσωπικότητας των ατόπων, το δικαίωμα στην ασφάλεια, στην ε, πολιτική, την εκπαιδευτική, ε, στην ευθύνη που υπάρχει για την υποδοχή των ξένων και την πολιτική για τις τοπικές μεταφορές. Πολλά από τα δικαιώματα που αναφέρει η χάρτα αφορούν θέματα γενικής φύσεως που αφορούν διάφορους δημόσιους φορείς. Τα δικαιώματα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αναπήρων κτλ. Σε ό,τι αφορά τα, ε, τα δικαιώματα που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια σε πολλά κράτη, οι διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με την άσκηση του δικαιώματος παραμονής, υποχρέωση εγγραφής ε, στους καταλόγους των ε, αρχών όπου κατοικεί κανείς. Αυτά όλα τα θέματα είναι αρμοδιότητα των τοπικών αρχών. Ο, ο Ευρωπαίος πολίτης που θέλει να διαμείνει στην Ιταλία πάνω από τρει μήνες θα πρέπει να εγγραφεί στο, στην κοινότητά του, ε, όπου διαμένει, στην κοινότητα που διαμένει. Η ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών ξεπερνάει τις απλές διατυπώσεις διοικητικής φύσεως. Ο... Και έχουν ένα ρόλο πολύ σημαντικό σε σχέση με την πολιτική υποδοχή των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, ό,τι αφορά την, ε, την, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, ε, τη στέγη κτλ. έχουν και εκεί σημαντική ευθύνη. Με βάση όλα αυτά είναι σαφές ότι η ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων που αναφέρει ο χάρτης είναι μια διαδικασία που σημαίνει δράσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στο διεθνές, στο ευρωπαϊκό, στο κρατικό, αλλά και στο περιφερειακό και στο τοπικό, στην τελική ανάλυση. Αυτό έχει υποθεί πολλές φορές από την Επιτροπή των Περιφερειών και αναγνωρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδίω στο ψήφισμα της 14ης Ιανουαρίου 2009 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2008. Αυτό το ψήφισμα υπογραμμίζει το ρόλο που οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να παίξουν για την εφαρμογή και την προώθηση αυτών των δικαιωμάτων. Η σημασία της συνεργασίας των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Φερρυπίν, όταν ας πούμε, η συλλογή των δεδομένων και των καλών πρακτικών υπάρχει, και μέσω του διαλόγου ε, της Επιτροπής ε, ΣΥΒΕΞ, της Επιτροπής των Περιφερειών δηλαδή, για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα. Παρά όλα αυτά τα προφανή που σας ανέφερα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων, αυτές οι λειτουργίες, αυτές οι αρμοδιότητες δεν αναγνωρίζονται ρητά. Δεν μπορούμε δηλαδή παρά να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε, γύρω από το οποίο σήμερα γίνεται όλη η συζήτηση, δηλαδή την έκθεση 2010 για την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή των Περιφερειών συζητάει αυτή τη στιγμή μια γνωμοδότηση για τη στρατηγική, ε, για την πραγματική ενεργοποίηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Άκανσον και ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά της. Εκεί εκφράζουμε σοβαρές επιφυλάξεις. Η έκθεση του 2010 για την εφαρμογή του χάρτη μιλά για την ανάγκη να ενημερώνεται καλύτερα τα άτομα για το πεδίο εφαρμογής του χάρτη και για τον τρόπο να εξασφαλίσουμε τα, το σεβασμό των δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβίασης. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, παρεξηγήσεις. Ε, αυτό φαίνεται από τον αριθμό των καταγγελιών των ε, φυσικών προσώπων προς την Κομισιόν και που αφορούν ε, τις συμπεριφορές κρατικών οργάνων που δεν εντάσσονται όμως στο πεδίο εφαρμογή του χάρτη. Από την άλλη, υπάρχει ανάγκη να δώσουμε σε αυτούς τους πολίτες μια απάντηση ε, και να τους κατευθύνουμε ε, στη σωστή πόρτα για να ξέρουν πού μπορούν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους. Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών για αυτές τις δραστηριότητε ενημέρωσης για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο χάρτης και ο προσανατολισμός των θυμάτων είναι πολύ σημαντικός. Είναι πολύ κοντά στους πολίτες και βρίσκονται παντού, σε όλη την ε, επικράτεια των κρατών μελών. Οι τοπικές λοιπόν και περιφερειακές αρχές μπορούν να παίξουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το ρόλο ε, του μοχλού ε, πληροφοριών. Ε, χωρίς να μπορούν να δώσουν πραγματικά πολλές πληροφορίες στους, στους πολίτες. και εμείς μπορούμε να ενημερώσουμε τα υπόλοιπα όργανα ε, για τον τρόπο ε, που εφαρμόζεται ο χάρτης, όπως μας λένε οι πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς υπάρχουν γενικά φορείς και οργανισμοί ενημέρωσης ε, των πολιτών και παροχής βοήθειας προς τον πολίτη. Παραδείγματο χάρη, ο συνήγορος του πολίτη, ο οργανισμός για τις ίδιες ευκαιρίες, για το γραφείο των ξένων. Πρόκειται για φορείς όπου τα άτομα μπορούν να απευθυνθούν ε, καταρχήν ε, σε ένα πρώτο επίπεδο για το σεβάσμα των δικαιωμάτων τους. Μέσω συγκεκριμένων προτάσεων η Κομισιόν μπορεί να δρομολογήσει κάποιες πρωτοβουλίες για την κατάρτιση πρωτοβουλίου ε, προσωπικού που θα ε, δουλεύει σε αυτούς τους οργανισμούς και που ανήκουν στις τοπικές αρχές. Ε, να τους καταρτήσουν για, την, για το χάρτη το, που εφαρμόζεται και σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται όμως ο χάρτης. Μπορούμε επίσης να υπάρξει ένα άτομο το οποίο θα βοηθάει σε κάθε τέτοιο γραφείο ε, μία ας πούμε πύλη προς την οποία θα, θα απευθύνονται οι πολίτες. Το Europe Direct που υπάρχει επίσης παντού ε, μέσω γραφείων ε, που ανήκουν σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, θα πρέπει και αυτό να μπορεί να παίξει σημαντικό κεντρικό ρόλο και στην, σε επίπεδο ενημέρωσης αυτού του προσωπικού, κατάρτιση αυτού του προσωπικού, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης και τα Πανεπιστήμια. Και με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθεί πραγματικά ο πολίτης ή θα μπορούσαμε επίσης αυτό το μάθημα που γίνεται προς τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, τους δικηγόρους και τους δικαστές, το μάθημα που λέγεται Ρόμπερτ Σούμαν, θα μπορούσαμε να το επικαιροποιήσουμε ε, και να εντάξουμε εκεί και τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, Υπάρχει πρόσφατη πρωτοβουλία της Κομισιόν, ε, μιας ομάδας εργασίας, ε, Europe Direct, ε, που ενεργοποιείται στην Ιταλία και ετοιμάζει προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Τέλος, όπως έχει υποθεί πολλές φορές από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και από την Επιτροπή των Περιφερειών, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να υπάρξει μια κατάρτιση των μαθητών για τον χάρτη. Έχουμε πολύ θετικές εμπειρίες. Το 2008-2009 ε, στην περιοχή μου, στην Εμίλια Ρωμάνια, κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια στα σχολεία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επίσης η πρόταση για τα συγκεκριμένα σχέδια επικοινωνίας ε, με τα παιδιά. Είμαι πρόεδρος της ε, επαρχίας Ρέτζο Εμίλια, που έχει μια θαυμάσια εμπειρία και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να εγκρίνουμε μαθήματα κατάρτισης και υλικό ε, παιδαγωγικό, πολύ συγκεκριμένο, για να μιλήσουμε στα παιδιά και να μιλήσουμε και στους δασκάλους τους. Θα ήθελα να κλείσω τώρα, αναφερόμενοι σε ένα βασικό πρόβλημα που έχει τεθεί εδώ. Ε, και που το επισημαίνουμε και εμείς. Ποιο είναι αυτό. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι καρπός 70 ε, ετών ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κράτους Ευημερίας σε μία περίοδο ειρήνης στην Ευρώπη, με εξαίρεση την ε, θλιβερή ιστορία την πρόσφατη των Βαλκανίων και μια περίοδο όπου υπήρχε οικονομική ανάπτυξη, δημόσιες ανα... Ε, ταπάνες και βελτίωση της γενικής ευημερίας. Δεν ξέρω τα επόμενα 70 χρόνια πώς θα είναι. Ε, θα λοιπόν, πάνε καλύτερα. Αλλά θεωρώ ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά και θα αλλάξουν πολλά πράγματα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και τη δική μου, αλλά και εν γέννη στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα θέμα ε, να, να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να σκεφτούμε πώς τα θεμελιώδη δικαιώματα του χάρτη πώς θα τα προστατευτούμε, πώς θα, προστατε... πώς θα προστατεύσουμε αυτά τα νέα δικαιώματα απέναντι στην οικονομική κρίση. Τι προτεραιότητες θα πρέπει να έχουμε, με τι πόρους θα πρέπει να τις προωθήσουμε. Πώς θα αναδιοργανώσουμε τα κράτη μας και το κράτος ευημερίας που είχαμε μέχρι στιγμής όλα αυτά τα θέματα ε, θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Μαζί νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε νέες απαντήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και δύναμη και γνώση για να βρούμε την καλύτερη απάντηση και για να υπερασπιστούμε αυτή τη δημοκρατία που μπορεί να έχει και διαφορετικές αποχρώσεις σε σχέση με αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση και τώρα θα δούμε τώρα τι θα τι έχει να μας πει ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαίου Δημοσιολόγου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το επίκεντρο της συνεδρίας, το βασικό μας θέμα είναι η συνεργασία στο χειρισμό καταγγελιών για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ειδικότερα η συνεργασία μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού επίπεδου. Αν μου επιτρέπετε, στα δύο από τα δέκα λεπτά που μου δώσατε θα εξετάσω το θέμα της προηγούμενης συνεδρίας γιατί μέρος του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ένα κύριο κομμάτι του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να ασχολείται με καταγγελίες κατά των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, δίνει στους πολίτες και στους διαμένοντες στην Ένωση το δικαίωμα να ε, προσφύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για κακοδιοίκηση στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Η μόνη εξαίρεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης είναι το δικαστήριο ε, με τον ε, δικαστικό του ρόλο. Ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες κατά των αρχών στα κράτη-μέλη, αλλά όπως θα εξηγήσω, οι εθνικοί και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές μπορούν. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής Αναφορών αυτής της Επιτροπής, ο διαμεσολαβητής πάντοτε θεωρούσε ότι η κακοδιοίκηση περιλαμβάνει την αποτυχία να ε, τύχουν σεβασμού τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν ε, για πρώτη φορά ε, ανακηρύχθηκε ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2000, ο διαμεσολαβητής αμέσως άρχισε να τον εφαρμόζει στις ερευνές του. Επίσης, ε, αναλάβαμε έναν αριθμό πρωτοβουλειών με βάση το χάρτη, για παράδειγμα, την, ε, τις διακρίσεις ε, βάσει της ηλικία και τις διακρίσεις και την ελευθερία έκφρασης των υπαλλήλων. Τώρα που ο χάρτης έχει την ίδια νομική αξία όπως οι συνθήκες, συστηματικά τον λαμβάνουμε υπόψη το χάρτη στις ερευνές μας ακόμα όταν βέβαια έχει νόημα αυτό, ακόμα και αν δεν επικαλείται η ίδια η καταγγελία το χάρτη. Ε, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία να δώσω, αλλά είναι υψηλό ποσοστό των καταγγελιών στα πλαίσια της ε, εντολής μας αφορούν στον χάρτη. Οι βασικές διατάξεις ε, έχουν να κάνουν με τις μη διακρίσεις, το περιβάλλον, την πρόσβαση στα έγγραφα και βέβαια την καλή διοίκηση, πράγμα που εγγυάται 41 του χάρτη. Όμως, οι περισσότερες καταγγελίες που αφορούν τα δικαιώματα ε, που απορρέουν από το χάρτη δεν εμπίπτουν στην ε, δική μας εντολή επειδή ε, στρέφονται κατά των αρχών των κρατών μελών οι διαμεσολαβητές που έχουν την εντολή να ασχολούνται με τέτοιε ε, προσφυγές είναι οι εθνικοί και περιφερειακοί διαμεσολαβητές στα κράτη-μέλη. Και ο Ευρωπαίο διαμεσολαβητής είτε ε, μετα... διαβιβάζει αυτές τις ε, καταγγελίες ή συμβουλεύει τους προσφεύγοντε που να απευθυνθούν. Έτσι πρέπει να είναι η επικουρικότητα στη διοίκηση, στην απονομή του δικαίου της Ένωσης και και τη διοίκηση της πολιτικής ε, συνοδεύεται από επικουρικότητα στα ένδικα μέσα. Γι' αυτό ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και οι διαμεσολαβητές στα κράτη-μέλη έχουν ένα δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Διαμεσολαβητών, που μας βοηθάει να εξυπηρετούμε συλλογικά καλύτερα τους πολίτες. Η συνεργασία στο δίκτυο στηρίζεται σε δύο πτυχές. Το πρώτο είναι να διασφαλίσουμε ότι οι καταγγελίες θα πάνε στον αρμόδιο διαμεσολαβητή το ταχύτερο δυνατό και το δεύτερο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε κάθε θεσμικό όργανο να μπορεί να ε, είναι αποτελεσματικό στην εντολή του ε, Μπορεί ο εθνικός και ο περιφερειακός διαμεσολαβητής να ρωτήσουν τον Ευρωπαίο ε, διαμεσολαβητή σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία και την ερμηνεία της και το χειρισμό συγκεκριμένων ε, καταγγελιών. Οι ε, απαντήσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά μπορεί να βοηθήσουν τον διαμεσολαβητή που ερωτά να διαμορφώσει άποψη. Πολλές ερωτήσεις τις προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της μας βοηθάει να διατυπώσουμε τη σωστή απάντηση στον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή. Δηλαδή σε ενωσιακό επίπεδο συνεργαζόμεθα και με την Κομισιόν για να βοηθήσουμε τον εθνικό διαμεσολαβητή να ερμηνεύσει θέματα ενωσιακής νομοθεσίας που προκύπτουν στις έρευνές τους. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία έρευνα που να αφορά στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων η εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι οι εθνικοί διαμεσολαβητέ είναι πιο έμπειροι σε υποθέσεις που θέτουν θέματα ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στα πλαίσια του Εθνικού του Συντάγματος ή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ας πούμε σε θέματα της κοινή αγροτικής πολιτικής που είχαμε ε, υποθέσεις. Έτσι περνώ στο βασικό θέμα μου σήμερα αυτό που ανέφερε σήμερα το πρωί η Επίτροπος Ρέντινγκ στην ε, παρέμβασή της. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν, αφορούν συγκεκριμένες καταστάσεις όπου ο προσφεύγων θεωρεί ότι έχει αντιμετωπιστεί ε, δυσμενός και θέλει αποκατάσταση. Οι προσφεύγοντες αναφέρονται στο χάρτη γιατί ξέρουν ότι είναι ευρωπαϊκό, ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφεύγουν σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επιτοπλίστων όμως θέλουν απλώς ε, αποκατάσταση. Δεν τους ενδιαφέρει που θα στηριχθούν στην ομολογία, στη σύμβαση, στο χάρτη, στην σύμβαση του άρχους, τη σύμβαση των, του, των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Δεν τους ενδιαφέρει που θα στηριχθούν. Θέλουν όμως επανόρθωση, αποκατάσταση. Τώρα αυτό τι σημαίνει για την πολιτική μας. Ε, θεωρώ ότι η πρώτη επίπτωση αφορά την γνώση του χάρτη από την κοινή γνώμη. Η καλύτερη ε, ενημέρωση είναι σημαντικός ε, στόχος. Υπάρχει μια μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε μια έρευνα ε, στην αρχή του χρόνου και οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες είπαν ότι θεωρούν ότι το πιο σημαντικό καθήκον του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή είναι να τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους. Και αυτό είναι ένα έβριμα που το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Και προβληματιζόμαστε εσωτερικά, ας πούμε, πώς θα απαντήσουμε σε αυτό και πώς θα συνεργαστούμε με την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να δώσουμε συνέχεια σε αυτά τα ευρήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζει ο κόσμος περισσότερα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε και θα απογοητευτούμε αν περιμένουμε ότι έτσι θα μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών που επικαλούνται το χάρτη ενώ αυτός δεν εφαρμόζεται. Η δεύτερη ε, πίπτωση αφορά μια αρχή που ανέφερα προηγουμένως. Η επικουρικότητα στα ένδικα μέσα. Ουσιαστικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δέχεται πολλές καταγγελίες κατά των εθνικών αρχών. Όπως εξήγησα, αυτές τις διαβιβάζουμε στον αρμόδιο διαμεσολαβητή στο δίκτυο ή συμβουλεύουμε τον προσφεύγοντα να απευθυνθεί σε εκείνον τον διαμεσολαβητή. Εκ μπορώ να πω ότι αυτός είναι κατ' ουσίαν ένας μονόδρομος. Σπάνια ένας εθνικός διαμεσολαβητής μεταβιβάζει μία, διαβιβάζει συγγνώμη, μία καταγγελία στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Γιατί, διότι δεν λαμβάνουν καταγγελίες που να, απευθύνουν, που να τάσσονται κατά της διοίκησης της Ένωσης και όχι κατά της εθνικής διοίκησής τους. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο, θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση αν το πρώτο ενστικτοδός πρωτίστως οι προσφεύγοντες πήγαιναν στον εθνικό και όχι στον Ευρωπαίο ε, διαμεσολαβητή, ούτως ώστε ο εθνικός διαμεσολαβητής να στέλνει υποθέσεις σε εμάς και όχι αντίστροφα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει μια νυχτή. Δεν θα χρειάζονταν όμως ε, νομοθετικές αλλαγές για να γίνει αυτό το πράγμα ή να αρχίσει να γίνεται. Είναι θέμα ε, στάσης της κοινή γνώμης μέσα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ε, Δίκτυο Διαμεσολαβητών εμείς ε, αρχίσαμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος του κάθε διαμεσολαβητή και να είναι γνωστό. Κάναμε και μια δήλωση ε, που αναφέρεται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και, στα, και στους διαμεσολαβητές ε, μπορέσαμε έτσι να αυξήσουμε την ορατότητα του δικτύου στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε ένα λογότυπο για το δίκτυο για να το μαθαίνει ο κόσμος και έχουμε και έναν διαδραστικό οδηγό για να βοηθάμε τους ε, προσφεύγοντες. Σε δύο εβδομάδες δε Ό οι εθνικοί διαμεσολαβητές στο δίκτυο θα συναντηθούν στην Κοπενχάγη. Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση θα είναι η ανάπτυξη του δικτύου και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ, του κενού τέλος πάντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών. Μέρος του κενού που πρέπει να πληρώσουμε είναι αυτό ότι ο χάρτης πολλές φορές θεωρείται κάτι για το οποίο πρέπει να πάμε στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο για να έχουμε επιτυχία. Αυτό που πρέπει να στοχεύσουμε είναι μια κατάσταση όπου θα νιώθουν εμπιστοσύνη οι ενδιαφερόμενοι και δικαίως ότι υπάρχει ένα ανεξάρτητος φορέας αμερόληπτος στη χώρα τους που θα τους βοηθήσει να βρουν το δίκαιο τους και όπως αυτό ενδεχομένως μπορεί να απορρέει από το χάρτη, όταν, εάν εφαρμόζει το χάρτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Και τώρα δίνω το λόγο στον καθηγητή Άλαν Μίλλερ, ο οποίος είναι πρόεδρος τη Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σκωτία και πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Ομάδας Εθνικών Θεσμών για τα, Ευρωπαϊκά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Και Δήμων, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με προσεκάλεσε ούτως ώστε να μπορέσουμε να το τοποθετηθούμε και εμείς στη σημερινή εκδήλωση. Να μην παρά αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι από τους άλλους φορείς για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος και είμαστε το τελευταίο πάνελ, οπότε θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντομος. Θε να τα πω γίνεται πιο απλά και λακωνικά, αλλά και το κάνω και ακόμα και τον πιέζει χρόνο, οπότε θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι γίνεται με αυτή την, την συνυπευθυνότητα, αυτό το οποίο ανέπτυξε η, κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπο σήμερα το πρωί. Και οπότε θα πρέπει να δούμε ευρύτερα το θέμα αυτό τη συνυπευθυνότητα. Πρώτα πρώτα. Θα σας πω ότι οι αξίες που προωθεί ο Χάρτη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για θεμελιώδη έξι Ευρωπαϊκή Ένωση. όμω όμως, όμως, εγώ θα ήθελα να σα προτρέψω να το δούμε το θέμα ευρύτερα. Να δούμε δηλαδή <clears throat> και την ερμηνεία και τον ε, δυνάμει ρόλο του, του χάρτη πέρα από τι δυνατότητε τη στενάτη και την ε, εφαρμογή. Ευρύτερη προσέγγιση σημαίνει ότι ε, πρέπει να καταλάβει κανεί τον χάρτη και αυτό είναι μέρος Ενό πλαισίου για προστασία, για ευθύνε των κρατών, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Συμβουλή τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο, το προβλέπει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και επίση αυτά προβλέπονται ε, λόγω του ότι έχει προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την προσχώρηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Σύμβαση. Έχουμε κυρώσει δε όλε τι συμφωνίε που προβλέπουν τι υποχρεώσει ε, που απορρέουν από τον ΟΗΕ. Οπότε τα περισσότερα που σου ακούστηκαν σήμερα που ήταν τόσο ενδιαφέροντα για μια που ανταλλάξαμε γνώσει, ιδέε, εμπειρίε, άκουσα σήμερα επανειλημμένα το πώ μπορούμε να καλύψουμε το πρόβλημα του να πηγαίνουν τα φυσικά πρόσωπα να χτυπούν τη λάθος πόρτα. Επομένως, αυτή η ευρύτερη προσέγγιση μας βοηθά και σε αυτό το πρόβλημα. Μας κάνει να είμαστε ίσως πιο αποτελεσματικούς. Διότι, για παράδειγμα, ευρύτερη προσέγγιση προς τον ε, χάρτη, την ερμηνεία του, την εφαρμογή του, τη σημασία του σημαίνει ότι ίσως δεν πρόκειται τελικά περί λάθο, όταν κανείς χτυπάει λάθο πόρτα. Όταν κανεί την αξιοποιήσει το χαρτί, γιατί όλοι θα ξέρουμε, αυτό το οποίο είπε ο κύριο ή η κυρία Γκίλη, καθηγήτρια με το πρωί, σε σχέση με, με τα ελληνοτουρκικά σύνορα, σε σχέση με τη, με τη Frontex, σε σχέση με τι συνθήκε κράτηση. Και ε, πάρα πολύ θετικό είναι αυτό το οποίο είπε ο Ιάννη προηγουμένω, ότι αυτό το θέμα θα το εξετάσει ο διαμεσολαβητή. Πάντω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι αυτό δεν είναι θέμα του χάρτη. Πάντως, αυτή η ευρύτερη προσέγγιση τι σημαίνει. Ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνούν τις, ε, ε, τις, τις ε, υποχρεώσεις τους δυνάμει της Σύμβασης των Δικαιωμάτων σε σχέση με το, όταν ενεργούν ως μέλη στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κρατημέλη έχουν βασικό καθήκον να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΟΗΕ και από τη Σύμβαση γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι δυνατόν κανείς να έχει μια μπακάλικη προσέγγιση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρωπίνα δικαιώματα πρέπει να διαπνέουν πάσα πολιτική. Περιφερειακή, τοπική, διεθνή. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένα είδου στενόμυαλη και στενή ερμηνεία και κατανόηση για τον χάρτη. Ευρεία προσέγγιση και έτσι κανείς αντιλαμβάνεται το πόσο ο χάρτης μπορεί να λειτουργήσει. Βεβαίως και υπάρχουν και θέματα διαδικασίας, θέματα δικονομικά, το πώς τέλος πάντων μπορεί ο κάθε φορά προσβαλόμενος να αποκατασταθεί και με, με, με το λιγότερο δυνατό μπελά. και ξέρουμε πόσες υποθέσεις εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, τι γίνεται με τα, με, τις, τα αιτήματα και καταγγελίες κλπ. Είναι και θέμα επικουρικότητας. Είναι θέμα υλοποίησης του χάρτη και της σύμβασης ανθρωπινών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Άρα, να, πώς προκύπτει η δύσκολη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, πώς προκύπτουν ε, οι καταγγελίες, πώς προκύπτει το πρόβλημα του να χτυπάει κανείς τη λάθος πόρτα. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα περισσότερο και ο συνάδελφος, η συνάδελφος Ντες Χόγκεν μίλησε προηγουμένως για τα website, για την ε, αλληλοενημέρωση, για την ε, κατεύθυνση των καταγγελιών στους κατάλληλους διάβλους. Όλα αυτά είναι κομμάτι της λύσης, είπαμε και τι κάνει και το Συμβούλιο της Ευρώπης και τι κάνει και το Δικαστήριο. Επίσης, για να δούμε πώς είναι το ευρύτερο τοπίο σε σχέση με τις καταγγελίες και τη διαχείρισή τους. Υπάρχει συμπευθυνότητα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και σήμερα αυτό που με εξέπληξαν ήταν κάποια σχόλια που ακούστηκαν σήμερα το πρωί και τα οποία απηχούσαν κάποιο, κάποιο θεμητό προβληματισμό όσον αφορά ακριβώς αυτά τα κέντρα κρατουμένων στην Ελλάδα και τα συστημικά προβλήματα που είναι η ρίζα του κακού. Ταυτόχρονα, για βρείτε την εικόνα, ποια είναι. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες αυτό έχει την τιμή του, αλλά το τίμημα το σχετικό θα πρέπει να καταβληθεί. Η απάνθρωπη μεταχείριση δεν είναι θέμα προπολογισμού, είναι ένα απόλυτο δικαίωμα. Επομένω, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να, να, να συμβαδίσει αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς με τα μέτρα λιτότητας της ελληνικής κυβέρνησης και, και θα πρέπει όταν συνοείται η Κομισιόν για τα μέτρα λιτότητας με την ελληνική κυβέρνηση βάζει το θέμα αυτό στο τραπέζι βλέπουν όταν γίνονται αυτές οι, αυτές οι, οι περικοπές έχει κάτι κανείς να εξετάσει βοηθάτε βοηθάτε η, η Ελλάδα να τηρήσει την υποχρεώσει, μια που έχουμε πλημμυρίδα καταγγελιών σε Βρυξέλλες και Στασβούργο είναι συνυπεύθυνοι όλοι. Δεν θα πρέπει με τα κράτη-μέλη να αφήνουν από την πόρτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι τρέχουσε υποχρεώσει του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρακτικέ προτάσει τώρα, εν κατακλείδη. Τι θα μπορούσε να απαιτεί αυτήν την συνυπευθυνότητα. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Ομάδα θα πρέπει να λειτουργούμε σαν γέφυρα. Γιατί έχουμε τις χώρες, τις εθνικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές. Άρα έτσι θα βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και τα κρατημέλια. Ούτως ώστε να θεσπίδεται σωστοί νόμοι, να ακολουθείτε σωστή πρακτική, και έτσι να εξασφαλίσουμε το πώ θα τηρούνται τα αρθροναδιό μα γιατί δεν υπάρχουν προσφυγέ, καταγγελίε και δικαστήρια. Το πιο, η πιο καλή ρύθμιση είναι η πρόληψη. Άρα, άρα ξεκινούμε από την νομοβαστική διαδικασία. Να τι θέλουμε να πετύχουμε. Και σε συνεργασία με διαμεσολαβητέ. Εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τι εκμεταλλευτεί. Τώρα όσον αφορά το τμήμα της υπευθυνότητας, της ευθύνης μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναγνωριστεί το πόσο αξίζει η πρωτοβουλία μας Πέρασα στην Τουρκία μερικές μέρες και από την Τουρκία θα κατευθύνει εδώ τώρα και παρακολούθησα την ε, Εθνοσυνέλευση Είδα τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό κράτο, συναντήθηκαμε και με οργανώσει, με αντισανομικού και αυτό το οποίο ήθελα ήταν να βοηθήσω να συγκροτηθούν κάποιοι φορεί για ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι έχει ε, δημιουργηθεί λόγω τη προσχώρηση στην Τουρκία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχει μεγάλη πρόοδος, ε, έχει ανέβει ο πύχη για την προστασία των δικαιωμάτων και επίσης ε, θα, θα, έφερνε μηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το να βρεθεί ενώπιον τη εξή καταστάσεω. Όσοι στην Τουρκία δεν είναι και τόσο φανατικοί για να έχουν ένα φόρο δικαιωμάτων και όμως δίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, για κοιτάξτε, λιγότερα από τα μισά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φορέα τα δρομένα δικαιώματα που αντιστοιχεί στα πρότυπα που έχει τάξει ο ΙΕ. Άρα εμείς η Τουρκία θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ λογικό, λογική αυτή η αξίωση. Δεν το λέω αυτό γιατί δεν χρειάζεται προσέγγιση με μας στην Τουρκία, αλλά σας το λέω ότι αυτό στριμώχνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτέ τις παγκοσμίες αξίες που λέμε ότι είμαστε παράδειγμα προ μήνυση. Όμως, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αναγνωρίσει το ότι θα πρέπει τα περισσότερα μέλη να λάβουν κάποια πρακτικά μέτρα ούτως ώστε τέτοιους οργανισμούς προστασία να τους ε, αναβαθμίσουν, να τους εγκροτήσουν. Να είχαμε εδώ κάποιο συνάδελφο από την, ε, από την ε, Ελληνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρετε, η Ελληνική Επιτροπή τι προπολογισμό έχει. Όχι πάνω από 100.000 ευρώ είναι αυτή η προκολότηση και ξέρουμε, ξέρουμε τι προκλήσει έχει αντιμετωπίσει σήμερα στην Ελλάδα Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και ακόμα και αυτές οι 100.000 προοικοδότηση κινδυνεύει λόγω των μέτρων λιτότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και να πιάνει είναι η συνυπευθυνότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την, για την Ευρωπαϊκή Ομάδα Οργανώσεων ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα, θα πρέπει η ομάδα μας να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Merci beaucoup pour... Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε που είναι τόσο δημιουργικά. Θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι και εμείς συμφωνούμε με το στόχο αυτό του να εμβαθύνουμε τον διάλογο για τις επαφές μας μεταξύ ε, αυτών των, ε, αυτής της ομάδας φορέων μεταξύ ημών και ημών τέλος πάντων. Και τώρα δώσουμε τώρα το λόγο στον επόμενο. Ο κύριος Καντάρ, Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων για την Ισότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση προς την Equinet να μιλήσει εδώ. Είναι ένα δίκτυο με 33 μέλη σε 88 χώρες. Στηριζόμεθα σε τρεις οδηγίες την... τρεις οδηγίες είναι πολύ ε, ειδική η θέση μας. Είμαστε μέλος, μέρος της δημόσιας διοίκησης, αλλά υποτίθεται ότι είμαστε ανεξάρτητοι και από την κοινωνία των πολιτών και από την κυβέρνηση. Ε, πώς λειτουργούν σύμφωνα με τις, ε, πώς λειτουργεί το Equinet ανεξάρτητη παροχή συμβουλών σε θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν πρόκειται για την εφαρμογή του χάρτη των οδηγιών της Ένωσης κλπ. Αλλά παίζουν ρόλο και στην ανταλλαγή πληροφοριών με τους ευρωπαϊκού φορείς και αυτό αναφέρεται ρητά σε μία από τις οδηγίες. Έχουν ρόλο να παίξουν λοιπόν διότι έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται με τους ευρωπαϊκούς φορείς ώστε να υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας. Επίσης ε, κάνουν και ε, έρευνες και διοργανώνουν και καμπάνιες και προάγουν ορθές πρακτικές, επίσης συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των μελών μας. Ε, υπάρχουν και επικαλύψεις ως ένα βαθμό και με τους ε, Εθνικά Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα εθνικά. Ορισμένα μέλη είναι μάλιστα τέτοια Εθνικά Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπάρχουν παραδείγματα και τάσεις ενδεχομένως όπως να τις πούμε ε, γιατί κάποια εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναλαμβάνουν μόνο να παίξουν ρόλο για την ίση μεταχείριση, τη διασφάλιση ίση μεταχείριση, αλλά γίνονται και ιδρύματα καθ' αυτά όπως στην ε, ε, Ολλανδία. Υπάρχουν ε, δύο διαφορετικοί φορείς τέτοιων φορέων ισότητας. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες διαφοροποιήσεις, αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς χειρίζονται τις καταγγελίες και τι κάνουν. Έχουμε φορείς που ε, είναι ιονοί δικαστικές αρχές και δέχονται καταγγελίες, άμεσα κάνουν έρευνες και τις χειρίζονται και αποφαίνονται. Και η απόφαση μπορεί να είναι να μην είναι νομικά δεσμευτική. Επίσης ε, προωθούν την ισότητα. Άλλοι έχουν ε, φορείς με λίγο διαφορετικό ρόλο. Ο βασικός ρόλος εδώ είναι η προαγωγή της ισότητας, καλές πρακτικές, αφύπνιση, ε, έρευνα και βεβαίως παροχή συμβουλών και υποστήριξη στα θύματα. Ε, αυτά κάνουν οι φορείς ε, ισότητας. Βέβαια κάποιες, κάποιοι φορείς που είναι οι ιονοί δικαστικές αρχές κάνουν και καμπάνιες ενημερωτικές και συμβουλεύουν για τις ορθές πρακτικές. Αυτό, αυτές είναι υπηρεσίες που παρέχονται σε εργοδότες και παρόχους υπηρεσιών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι σήμερα μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια προβλήματα στο ευρωπαϊκό σύστημα γιατί οι οδηγίες που ανέφερα ε, απαιτούν μόνο τη σύσταση εθνικών φορέων ισότητας για θέματα ε, φίλου, φιλής ε, και δεν ορίζουν ακριβώς την εντολή αυτών των φορέων. Οπότε υπάρχει εδώ κάποιο κενό στην νομοθεσία και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και αν πολλά κράτη-μέλη πάνε ένα βήμα παραπέρα και παρέχουν μεγαλύτερα επίπεδα προστασίας, υψηλότερα. Βεβαίως και αυτό συνδέεται με αυτό που είπε και ο Άλαν Μίλλερ, το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και απασχολεί πολύ τους φορείς ισότητας και τα ιδρύματα τα εθνικά για τα θεμελιώδη δικαιώματα και χρειαζόμαστε, πιστεύομαι, νομικά δεσμευτικά πρότυπα ώστε οι φορείς ισότητας να μπορούν να στηρίζονται ε, σε αυτά για να εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ανεξαρτησίας, λειτουργικά πρότυπα, δημοσιονομικά πρότυπα ε, που πρέπει να τα έχουν οι φορείς ισότητας ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να παρέχουν, όπως είπαμε, επαρκές επίπεδο προστασίας στους πολίτες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Μπάτλερ από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και άλλοι το είπαν ε, είναι το θέμα των προβληματικών εκθέσεων. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουν τι κάνουν οι θεφορείς, οι πολίτες για να χτυπήσουν τη σωστή πόρτα. Και αυτό δεν υπάρχει Οπότε πράγματι συμφωνούμε με τη διαπίστωση που έγινε. Γνωρίζουμε από την έρευνα ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει για τους φορείς ισότητας και όχι μόνο. Γενικά δεν γνωρίζουν τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Οπότε δεν γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους, δεν έχουν κουλτούρα προάσπιση δικαιωμάτων και να τα γνωρίζουν ακόμα είναι απρόθυμοι να πάνε είτε γιατί δεν εμπιστεύονται το σύστημα και τις δημόσιες αρχές ή δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά θα φέρουν κάποια αλλαγή. Και βεβαίω υπάρχουν και άλλες δυσκολίες όταν πρόκειται για ευάλωτε ομάδες όπως τους φιλομεταβατικού ή του Ρωμά. Το Equinet έχει πολλές δραστηριότητες εμείς όμως δεν είμαστε μηχανισμός ε, καταγγελιών. Ε, έχουμε μία μικρή γραμματεία εδώ στις Βρυξέλλες και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ε, ικανότητα των μελών μας ώστε να μπορούν να χειρίζονται αυτές τις καταγγελίες για διακρίσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε ειδικευμένους, έχουμε δραστηριότητες μέσα σε ομάδες εργασίας, που εστιάζουν στις επικοινωνιακές δραστηριότητες που μπορεί να έχουν οι φορείς ισότητας για να ενημερώνουν τους πολίτες ε, για τις δυνατότητες που έχουν και που μπορούν να προσφύγουν. Και το είπαμε αυτό πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ε, ότι δηλαδή ο κόσμος δεν έχει την πληροφορία. Πρώτα χρειάζεται να πάρει την πληροφορία και μετά ίσως αρχίσουν να εμπιστεύονται περισσότερο το σύστημα και να έρχονται σε εμά και να αρχίζουν να ε, καταθέτουν τις καταγγελίες τους. Το Equinet βέβαια προτίθεται και το κάνει, συνεργάζεται δηλαδή με όλους τους ε, Ευρωπαϊ, Ευρωπαίους εμπλεκομένους, ε, θεσμικά όργανα, ε, το Συμβουλίο της Ευρώπης, το, την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Εθνικών Φορέων, κοινωνικούς εταίρους, κοινωνία των πολιτών κλπ. Και είμαστε ευτυχείς γιατί ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να συνεργάζονται με όλους τους εθνικούς εμπλεκομένους σε εθνικό επίπεδο και αυτό γίνεται. Και αυτή η συνεργασία σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι οδηγεί σε μια πιο καθαρή κατανόηση των ε, δυνατοτήτων και των εντολών των διαφόρων ε, δρόντων και των μηχανισμών προσφυγής και αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνουν οι διάφοροι φορείς για τον πολίτη. Και σε τελευταία ανάλυση αυτό οδηγεί σε πιο καλή ε, λειτουργία του συστήματος ε, της διαβιβάσεις υποθέσεων αλλού, γιατί ε, οι δομές συνεργασίας, οι φορείς, οι οργανώσεις, καμιά φορά δεν ξέρουν και μεταξύ τους τι κάνουν, δηλαδή τι εντολή έχουν οι άλλοι. Οπότε πολλές φορές πρέπει να το συζητήσουν το θέμα για να δουν τι κάνει ακριβώς ο άλλος φορέας και τότε θα μπορέσουν να διαβιβάσουν ή να ε, στείλουν τις υποθέσεις που παραλαμβάνουν στους καθήλυν αρμόδιους οργανισμούς, αν εκείνοι δεν μπορούν να το χειριστούν το θέμα. Τέλος, ε, να πω ότι το Equinet ε, επίσης, η γραμματεία του Equinet δέχεται κάποιες λίγες καταγγελίες για τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και επειδή δεν μπορούμε να τα χειριστούμε αυτά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε και να αναπροσανατολίζουμε τους προσφεύγοντες στην αρμόδια εθνική ή διεθνή αρχή αν χρειαστεί η φορέα. Αυτά συνοψίζουν το έργο της Equinet, του Equinet, γιατί είμαστε μια πύλη προς όλους τους εθνικούς φορείς ισότητας και αυτό το κάνουμε για τα άτομα που έρχονται με καταγγελίες, το κάνουμε επίσης και ε, για θεσμικά όργανα της Ένωσης και όλους τους εταίρους μας, ούτω ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και να φτάνουν τους φορείς ισότητας. Προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας για την εφαρμογή του χάρτη. Χρειάζονται όλοι και οι φορείς στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα Εθνικά Ιδρύματα ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει, έχουν οι συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. να ονομάζομαι και κυρίως γραμματέας των φιλελευθέρων σε Μητρό Περιφερειών. Αλλά συμμετέχω και ηγούμε κάποιο μικρού κόμματο στην Ισπανία και θα ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Χάντι. Μας είπε και είναι κατανοητό ότι θα ήθελε οι πολίτες να προσφεύγουν καταρχήν σε εθνικούς φορείς πριν έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκά όργανα. Κάτι το οποίο βεβαίω είναι πρόβλημα παρουσίαση, είναι θέμα αντίληψη. Υπάρχει όμω εδώ πέρα κάτι το οποίο δεν το λάβατε υπόψη νομίζω. Διότι ε, ένα ε, βασικό λόγο. γιατί, τουλάχιστον στην Ισπανία, πολλοί ε, πηγαίνουν ε, πρώτα στις ε, θεσμικά όργανα είναι ότι δεν εμπιστεύονται ε, τις, εθνικές αρχές. Και αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους γλωσσικούς ή μπορεί διότι έχουμε ε, ξένους που έχουν έρθει από άλλη χώρα επειδή είναι βραδία η απονομή δικαιοσύνη ή διότι απλώς μπορεί να έχουμε αδύναμο το εθνικό Όταν Τώρα έχουμε, υπάρχει ένας περιφερειακός ο οποίος λένε για πολιτικούς λόγους ε, καταργείται. Οπότε, εντάξει, δεν είπα ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πλευράς περιφερειακής για να εξασφαλίσετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε, συγγνώμη, σε, εθνικό επίπεδο, να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη προς εθνικούς θεσμούς. Όμως, όσο συνεχίζονται αυτοί οι λόγοι που είπα και εσείς θα συνεχίζετε να λαμβάνετε ε, καταγγελίες από ε, τον κόσμο ότι εσείς πριν ο κόσμος προσφύγει εις εθνικές αρχές. Επόμενος. Ο επόμενος. Εγώ εκπροσωπώ την πρόεδρο του Ισπανικού Φορέα των ε, προσώπων που έχουν φυγεί από τον νόμο αυτόν για την περιουσία στην, στην παραλία της Ισπανίας, εχθές Ισπανίας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή εκδήλωση και θέλω να σας πω ότι αν δεν κάνω λάθος η αίσθηση που έχω είναι ότι ότι μας εξηγείται πως οι ευρωπαϊκές αρχές δεν θα μας βοηθήσετε εμάς που μένουμε στην Ισπανία εμάς, τους Ευρωπαίους Ισπανούς και μη Ισπανούς γιατί είμαστε πάρα πολύ που εκεί κατοικούμε πέστε μου παρακαλώ το δικαίωμα στην ε, ε ιδιοκτησία δεν είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αναδρομική δε εφαρμογή νόμου δεν αντιβαίνει στις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Η δε κατάσχεση, απαλωτρίωση ε, ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε νόμιμα δεν έρει την ασφάλεια του δικαίου. Τόσες είναι οι οικογένειες που τους απαλωτριώσανε. Μαγαζί, σπίτι κλπ. Μιλούμε για για πράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν νόμιμα. Μιλούμε για νόμο που εφαρμόστηκε αναδρομικά. Αυτό δεν είναι, δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Τι συνθήκη Λισαβόνας υπογράψατε. Γιατί δεν είναι δεσμευτική, το λέει και στα αγγλικά. Why. Γιατί δεν υπογράψατε. Γιατί το κοινοτικό δίκαιο δεν προσαρμόζεται σε αυτή τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί, γιατί. Τι να την κάνουμε, τη συνθήκη. Τι τη θέλουμε. Τι θέλουμε το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων εάν μετά δεν καλούνται οι χώρες να συμμορφωθούν. Είμαστε ή δεν είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες στην Ισπανία. Να το παραπονώ μου. Και έχω την αίσθηση ότι ήρθα εδώ και εσείς μου λέτε να μην προσφεύγω στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πηγαίνω πρώτα στα ισπανικά. 15 χρόνια κράτησε ο δικαστικό αγώνα, τον οποίο έχασα στην Ισπανία. Γιατί το 98% των υποθέσεων σε σχέση με τη γνωστή υπόθεση των ακτών, όλε τις οι αγωγέ απορρίπτονται. Είναι ύποπτο αυτό. Είναι στρεβλός αυτός ο νόμος. Θα, πρέπει να πάτε να ζητήσετε εξηγήσει από την Ισπανία. Και εγώ δεν πήγα και ξαναπήγα σε επιτροπές αναφοράς, πάρα πολύ ευγενικά με σποδέχτηκαν, όμως τελικά η Ισπανική κυβέρνηση έγραψε τα παλιά του υποδήματα αυτές τις επιτροπές αναφορών. Αυτές οι αποφάσεις είναι έολες των δικαστήριων των Ισπανικών. Εμείς αποκτήσαμε νόμιμα την περιουσία μας. Είναι ύποπτο, δεν συμφωνείτε, ότι να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος αναδρομικός, α, απαλωτριώσεις χωρίς αποζημίωση. Ε, δεν αντιβαίνουν όλα αυτά στο κοινωτικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Merci. Euh, Άλλες παρεμβάσεις παρακαλώ. Συνεχίζω, μετά, συνεχίζω μετά από εκεί που σταμάτησε ο Άλαν. Όλα από τα σχόλια τα προσυπογράφω. Επίσης, συμφωνώ και με αυτά που είπε ο Τόμας για την ανεξαρτησία των ε, φορέων ποιότητας αυτός. Ναι, φορέων συγγνώμη ισότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει για να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε ο Άλαν. Καταρχάς ο αριθμός αυτών των φορέων στα κράτη-μέλη. Είτε δεν αρκούν, είτε είναι αδύναμοι. Δεν έχουν αρκετές αρμοδιότητες. Είναι η τελευταία τροχή Η Κομισιόν ετοιμάζεται να κάνει κάτι αντίστοιχο με τις αρχές των Παρισίων για τους φορείς αυτούς ε, για την ισότητα ή θεωρείτε ότι είναι κάτι χωριστό και επομένως θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες αρχές. Merci. S'il n'y a pas propose. Je souhaiterais euh, Να απαντήσω στην ε, παρέμβαση που έγινε για τον Λέιντε Κώστα, για τον ε, παράκτιο νόμο. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να καταλάβουμε καλύτερα faire πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, ώστε να αποκτήσουν σάκα και οστά τα δικαιώματα του χάρτη είναι μια ευθύνη που την έχουμε από κοινού. Είναι το πρόβλημα όλων μας και των εθνικών αρχών και των περιφερειακών αρχών και των ευρωπαϊκών αρχών. Όλα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν σεβόμενοι το θεσμικό πλαίσιο που καθήκη της Λισαβόνας, με σεβασμό των θεσμικών και νομικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη δίνει κάποιε αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει το διαχωρισμό αυτό να τον έχουμε υπόψη μα. Σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα διάλογο μεταξύ της, ε, του ευρωπαϊκού επίπεδου και του εθνικού επίπεδου για να καταλάβουμε καλύτερα τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την, πραγματι, την πραγματική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως περιλαμβάνονται στη χάρτα. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε Συγκεκριμένε περιπτώσεις. Θέλουμε να ξεκινήσουμε διάλογο για να βρούμε λύσεις ούτω ώστε να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία. Με σκοπό βέβαια τελικό να βοηθήσουμε τον πολίτη. Αυτός είναι ο στόχος σήμερα. Φυσικά υπάρχουν ε, περιπτώσεις δύσκολες από νομικής απόψεως. Όπως αυτή, αυτός ο νόμος, ο Λέιντε Κώστα, ο νόμος για τις παράκτες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το θεμελιώδες δικαίωμα στην περιουσία. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε απλώς με την δικαιοδοσία, με την αρμοδιότητα. Δεν ξέρω ποιο δικαστήριο, το, η Κομισιο... το δικαστήριο του Στρασβούργου, του Λουξεμβούργου, η Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών, το γεγονός ότι οποιοδήποτε από αυτούς ε, λέει ότι δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα θεμελιώδων δικαιωμάτων. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε την κατάσταση. Ε, ζούμε σε ένα κράτο δικαίου όπου υπάρχει επιμερισμό των αρμοδιοτήτων. Δεν μιλάω για τη δική σα περίπτωση, την ειδική. Αυτό τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και ένα τρόπο για να το λάβουμε υπόψη, τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και των ρόλων του ευρωπαϊκού επίπεδου του εθνικού επίπεδου, του περιφερειακού επίπεδου και του Συμβουλίου τη Ευρώπη, να δούμε πώ μπορούμε να συνεργαστούμε παρά να μείνουμε στο status ο καθένα να λέει «Α, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι του άλλου». Πρέπει να κάνουμε πραγματική δουλειά συνεργασία. για να ξεπεράσουμε τι καθαρόεμε νομικέ ή νομικίστικες εξηγήσει, με σκοπό να δώσουμε χείρα βοηθεία στον πολίτη. Euh, Ξεκινήσουμε διάλογο για να βελτιώσουμε την κατάσταση για τον πολίτη που έχει πρόβλημα με τα θεμελιώδη δικαιώματά του που δεν γίνονται σεβαστά. Να πω δύο λόγια ακόμα. Αυτό που ανακαλύψαμε ασχολούμενοι με διάφορες αναφορές Ιδίω εκεί όπου υπάρχουν ισχυρισμοί για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ότι ο κόσμος περιμένει πολύ περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτά που εμείς μπορούμε να δώσουμε. Πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν η Ευρώπη να είναι πιο δυνατή, ούτω ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στι ανησυχίε των πολιτών. Αλλά έχουμε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Με αυτή δουλεύουμε και βραχυπρόθεσμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όσο περισσότερο όμω εκφράζονται οι πολίτες για αυτά τα θέματα, τόσο πιο δυνατή θα γίνει η φωνή τους. Ούτω ώστε τελικά να υπάρξει μια κατάσταση όπου τα δικαιώματα θα ενεργοποιούνται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ισχυρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η Επιτροπή Αναφορών Πέρα από τους φορείς που υπάρχουν στο εθνικό επίπεδο, πέρα από τον αριθμό τους, πέρα από το τι κάνουν, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι απογοητεύουν τους πολίτες. Γι' αυτό στρέφονται προς εμάς. Ίσως έχουν πολλές προσδοκίες ή παράλογες προσδοκίες. Τουλάχιστον όμως όταν στρέφονται σε εμάς τους παίρνουν στα σοβαρά. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι οι νόμοι δεν ισχύουν και οι κανόνε δεν έχουν καμία σημασία. Δουλεύουμε μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό εμείς, μέσα από μια πολιτική διαδικασία, προσπαθούμε να επιλύσουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ερχόμαστε σε επαφή με τι εθνικές κυβερνήσεις, με τα Υπουργεία, με τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Χρησιμοποιώντας τους διαμεσολαβητέ τον εθνικό ή τον περιφερειακό κτλ. Με τη βοήθεια των εθνικών βουλευτών, που συμμετέχουν στι εθνικές ε, επιτροπές αναφορών για να βρούμε λύσεις. Μερικές φορές η διαδικασία είναι δύσκολη γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση. Αλλά δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε την ε, δέσμευση που έχει η Επιτροπή Αναφορών να κάνει αυτή την προσπάθεια. Η Ευρώπη σημαίνει κάτι για πολλού πολίτε. Και με το να λέμε, κοιτάξτε την εθνική αρμοδιότητα, νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα. Για να ενισχύσουμε λοιπόν τους δεσμούς μεταξύ των εκπροσώπων των ε, οργανώσεων, μεταξύ των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα το που ακούμε σήμερα, ακριβώς ε, αυτό το θέμα πρέπει να, να προωθήσουμε, τη συνεργασία. Παραδείγματος χάρη, ε, με τον Πολωνό διαμεσολαβητή Είχαμε μια συζήτηση. Γιατί, Γιατί εμείς ήρθαμε σε επαφή μαζί του για να προωθήσουμε τα, δικαίωμα, ε, τα δικαιώματα ομοφιλοφίλων, ανδρών και γυναικών, φιλομεταβατικών κτλ. Ε, χάρη στην προσπάθειά μα έγινε αυτή η συζήτηση. Παραδείγματο χάρη η Ομοσπονδία Τυφλών ήρθε αυτή τη βδομάδα στην Επιτροπή μα. Κοιτάξτε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για τι υποχρεώσει τη Ευρώπη προ ανθρώπου με αναπηρίε. Στάθηκαν προ εμά για να εξασφαλίσουν ότι θα κάνουμε κάτι για να, σεβαστούν τα, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους για πρόσβαση σε βιβλία κτλ. και εποπτικό υλικό. Ζητήσαμε κάποιον από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης να μας πει τι άποψη έχει. Δεν μας είπε τίποτα. Πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση όπου Θα πρέπει πια να αναλάβουν τις ευθύνες οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και να το βλέπουν αυτό οι πολίτες για τα θέματα του χάρτη. Θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτω ώστε να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών του πολίτη. Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν περισσότερη Ευρώπη, αλλά υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι προφανές και απόκειται σε εμά να κάνουμε προσπάθεια για να μειωθεί αυτή η έλλειψη. Και κάθε διαμεσολαβητή σε κάθε επίπεδο να κάνει περισσότερο, ούτω ώστε να βοηθήσει του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ, Δαβίδ. Ιαν, μπορεί να απαντήσει ερωτήσει που σου οι βουλευτέ και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της εμπιστοσύνης και είπα προς το τέλος της ομιλίας μου ότι αυτό που θα ήθελα είναι να νιώθουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι και μάλιστα να είναι δικαιολογημένη η εμπιστοσύνη τους για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων στη χώρα τους ε, στους οποίους θα απευθύνονται για να προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα. Εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιος. Εδώ ε, μιλώ για τους διαμεσολαβητές και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Όταν μιλάμε για αναφορές, ε, αυτό είναι διαφορετικό, είναι μια πολιτική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι άμεσα εκλεγμένο δημοκρατικό όργανο και βεβαίως ε, η διαδικασία σκοπό έχει να εξασφαλίσει τη δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ μιλώ για τον διαμεσολαβητή, που εκεί η λογική είναι λίγο διαφορετική. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δίκτυο που δημιουργήσαμε ε, ε, συμπεριλαμβάνει και πώς να σας το πω, ε, μια επιμερισμένη κουλτούρα, αν μια κοινή κουλτούρα. Ο κύριος Μποντής που ήρθε το πρωί, που δεν είναι εδώ ακόμα, δεν είναι πια εδώ, τον άκουσα σε μια στρογγυλή τράπεζα στη Γενέβη λίγες εβδομάδες πριν και τον ρώτησαν εκεί, σε σχέση με τις αρχές του Παρισιού, πώς μπορεί κανείς να είναι ανεξάρτητο αυτός όταν ορίζεται από τον πρόεδρο της ε, Δημοκρατίας και απάντησε και είπε γιατί υπάρχει ένα δικαίωμα αχαριστίας. Αχαριστίας. Η ανεξαρτησία δεν είναι αυτό που γράφει το κείμενο, είναι και το πνεύμα. Είναι μια κατάσταση μέσα στο μυαλό. Άκουσα τον Δανό διαμεσολαβητή δηλαδή, που είπε ότι ένας διαμεσολαβητής που δεν έχει σύγκρουση με την κυβέρνησή του ακόμα και με το κοινοβούλιο του μερικέ φορέ, δεν κάνει σωστά το έργο του, δεν κάνει σωστά το καθήκον του. Σωστό είναι αυτό. Το δικαίωμα λοιπόν τη αχαριστίας, με το να ε, συναντιόμαστε συχνά και να εκφράζουμε τέτοια αισθήματα, δημιουργούμε μια κοινή κουλτούρα για να δημιουργήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη που χρειάζεται. Ευχαριστώ. you. Και εγώ θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Είμαι λίγο πιο απεσιόδοξος από τον κύριο Χάρντεν. Το θέμα είναι πώς να περιμένουμε να δείχνουν εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους φορείς, αν δεν υπάρχει σαφής υποστήριξη από το δικό μας το επίπεδο. Όταν βλέπουν ότι κάποιες κυβερνήσεις δεν στηρίζουν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε εξασφαλίζουν κάποια προστασία. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να ε, εξοπλιστούν οι φορείς και να έχουν και μια ανεξαρτησία. για να είναι αξιόπιστοι στη βοήθεια που παρέχουν στα θύματα. και σε το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επίσης πολύ καλή πλατφόρμα για να σκέφτεται κανείς και λίγο ανεξάρτητα, όχι μόνο να ακολουθεί ένα μπούσουλα και να ε, μαθαίνει για τις ορθές πρακτικές από παντού. Πολλές συζητήσεις έχουμε κάνει για το πώς θα φτάσουμε στις ευάλωτες ομάδες, πώς θα βεβαιωθούμε ότι θα εμπιστεύονται τους φορείς ισότητας. Και υπάρχουν καλά παραδείγματα γιατί μπορεί να γίνει κάποια δομημένη συζήτηση με τους Ρωμά για παράδειγμα ή ε, μπορούν να συσταθούν γραφεία περιφερειακά και τοπικά για να μην χρειάζεται να πάνε πάντα στην πρωτεύουσα για να βρίσκουν το φορέα ισότητας εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Ε, ε, ce Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι είναι η αρχή αυτή που κάναμε σήμερα. Πρώτη φορά από ό,τι ξέρω. Οι εθνικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές βρίσκονται μαζί. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι διαφορετικοί φορείς που παρεμβαίνουν και μιλούν για τα θεμελιώδη δικαιώματα τελικά μας βοηθούν για να αναπτύξουμε μια κουλτούρα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για να βρούμε την διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο. Φυσικά καθυστερούμε, φυσικά θα θέλαμε να, πάει, να μπορούσαμε να πάμε πιο γρήγορα, αλλά το σεμινάριο αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε κοινά προβλήματα. Πρέπει να βρούμε μαζί λύσεις. Και κυρίως να υποφεληθούμε από την εμπειρία σας. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, θα συνεχίσουμε το διάλογο με την Επιτροπή Αναφορών, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Αυτή την ε, πολυεπίπεδη προσέγγιση, που είναι κάτι σημαντικό για να δημιουργηθεί μια καλή πολιτική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε τη διευθυνσή μας, τα στοιχεία μας. Μπορείτε να ξανάρθετε σε επαρφή μαζί μας μπορείτε να μας απευθύνετε ερωτήσεις και εμείς ούτως ή άλλως θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας γιατί σας χρειαζόμαστε.